Good morning. I think we may as well start with the first report, which is the face of female poverty in the European Union. Unfortunately, Κοιτάξτε, δεν θα έρθει ο Γαβριήλ, αλλά ο Θωμάς είναι εδώ. Ορίστε. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη εκ μέρου της Γαβριέλας που δεν μπορεί να παραστεί γιατί κάτι της συνέβη, είχε μια επίγουσα δουλειά να κάνει. Αλλά επειδή συνεργάστηκα στη σύνταξη της γνωμοδότησης και συνεργάστηκαν και οι δύο επιτροπές γυναικών και κοινωνική, μπορώ να σας πω ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ των συντονιστών των δύο επιτροπών και έτσι η Επιτροπή ΑΠΑΣΧ θα ασχοληθεί μόνο με τα γενικά θέματα ενώ η Επιτροπή ΓΙΝ με τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες. Στην τελευταία συνεδρία των συντονιστών 43 τροπολογίες είχαν απορριφθεί με, στη βάση αυτής της συμφωνίας, της κατανομής. Και όσοι δεν έχουν αποσύρει ακόμα τις ε, απαράδεκτες αυτές τροπολογίες να τις αποσύρουν αμέσως. Η διορία λήγει για τις γιν στα μέσα Σεπτεμβρίου. Έλυγε. Νομίζω ότι γενικά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πραγματική διαφωνία για την προετοιμασία αυτής της δρομοδότηση. Υπήρξε συμφωνία, έκθεση μάλλον, για την καταπολέμηση της ανέχειας και η κυρία Τσίμερα ασχολείται αυτή τη στιγμή με τους συμβιβασμούς. Σήμερα θα προσπαθήσει να τους ε, υποβάλει και σε όλους τους σκιώδεις και μέσα στη βδομάδα θα βρεθεί, θα λήξει η διαδικασία αυτή για τους συμβιβασμούς και στις 9 Νοεμβρίου θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Η συγγήτρια έχει μόνο δύο-τρεις τροπολογίες που απορρίπτει την 22 και την 34. που αποκλείει την φτώχεια των παιδών τη 42 για τρεις διαφορετικούς δίκτες ανέχειας που ζητιέται να καταργηθούν και την 51 που αφορά την παράγραφο 5 και τον θετικό ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνική πολιτική για διαγραφή προτείνει αυτή. Αυτές τις τροπολογίες δεν μπορεί να τις δεχθεί η κυρία Τσίμερ. Και υπάρχουν κι άλλες τρεις, οι 52 πάλι της κυρίας Μάισνερ. Μάισνερ. Που αναφέρεται στο πρώτο τμήμα ενός συμβιβασμού και την 35 και 36 για την ανέχεια των παιδών που θα συμπεριληφθούν και αυτές σε συμβιβασμό. έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 50% της ανέχειας των παιδών. Η κυρία Τσίμερ δυστυχώς λείπει, αλλά έχουν μιλήσει εξ ονόματός της, συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι καταπολέμησης της ανέχειας και των γυναικών. Οι τροπολογίες σχεδόν όλες για το ίδιο θέμα μιλούν εκτός από καμιά δυο που αναφέρθηκαν ήδη. Όταν γράφαμε τις τροπολογίες, να συντάσαμε τις τροπολογίες, δεν γνωρίζαμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη γυναίκα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, πολύ δύσκολο πράγμα. Και μας είπαν ότι και η ανέχεια των παιδών δεν έπρεπε να μας απασχολήσει. Τώρα μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα λέει. Ε, όλα αυτά μας δυσκολεύουν τη ζωή ως σκιώδης. Τη λέξη γυναίκα λοιπόν την έβγαλα από δύο-τρεις τροπολογίες μου ώστε να είναι πλέον αποδεκτές αλλά πρέπει να βρούμε συμβιβασμούς διότι πολλές από τις τροπολογίες όντως αναφέρονται στο ίδιο θέμα, στο ίδιο σημείο. Οι δικές μου τροπολογίες στοχεύουν στο να μην απλώς θρηνούμε για την ύπαρξη της γυναικείας ανέχειας αλλά να βρούμε λύσεις. Και έπειτα η 35 στη Γερμανία είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε όχι γενικότερα για ανέχεια αλλά για, την, για ολόκληρο δίκτυο ανεχείας. Δεν ξέρω αν στις άλλες χώρες το λέτε αυτό αλλά είναι φανερό ότι αν γεννηθεί ένα παιδί σε μια φτωχή οικογένεια όπου δεν εργάζεται κανείς, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι πολύ δύσκολο να βγουν από αυτόν τον φαύλο κύκλο που λέμε εμείς στη Γερμανία της ανεχίας. Ενώ το θέμα είναι πώς να βγούμε από αυτόν. Γενικά όμως αναμένω τους συμβιβασμούς. Ευχαριστώ κύριε Λόπε Φοντάνια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν και γενικά να πω ότι δεν νομίζω ότι οι σύντροφοι που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ή έχουν αντίρρηση θα, έχουμε, θα έχουν τελικά μεγάλο πρόβλημα για την ανέβρεση συμβασμού με αυτές τις τροπολογίες γιατί νομίζω θα ήταν καλό να έχουμε ένα ενιαίο ομόφωνο κείμενο. Πριν να αναφερθώ στις επίμαχες τροπολογίες θα έπρεπε να εκφράσω και την απορία μου για κάποιες τροπολογίες που έχουν χαρακτηριστεί μη αποδεκτές οι οποίες φαίνεται ότι δεν μπορούμε να τις καταθέσουμε στην Επιτροπή των Γυναικών. Δεν θα ήθελα βεβαίως να αφισβητήσω την αρμοδιότητα της Προεδρίας, όμως να πω ότι δεν κατανοώ ποιο είναι το κριτήριο που ακολουθήθηκε ιδιαίτερα για τις τροπολογίες 27, 30, 54, 59, 70 και 74 της πολιτικής μου Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί πήρα τις τροπολογίες οι οποίες μιλάνε για εργατικά δικαιώματα, για ανασφαλή εργασία και δεν καταλαβαίνω πως όταν μιλάμε για τις γυναίκες δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Δηλαδή όταν μιλάμε για τις γυναίκες δεν μπορούμε να μιλάμε για απασχόληση. Τότε αν δεν γίνεται αυτό θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η επιτροπή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να αποδεχτούμε την απόφαση του Προεδρείου. Απλά και μόνο ήθελα να εκφράσω την δυσφορία και τη διαφωνία μου. Όσον αφορά τώρα τις ε, πιο αμφίβολες τροπολογίες, τουλάχιστον νομίζω θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία σε αυτές. Αναφέρομαι στην παράγραφο 1 στο σημείο 2 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θεωρώ ότι θα ήταν καλό να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και προσωπικά θα ήμουν υπέρ του να υπερασπιστούμε μια αύξηση της πρικοδότησης του ταμείου αυτού εν ώψη δηλαδή της αύξησης της απασχολησιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γυναικών. Με το στόχο αυτό, όχι όμως ως κάλυψη κοινωνικής ε, πρόνοιας, κάτι το οποίο προέρχεται και από άλλα εργαλεία. Για την 53 διαφωνώ και για την 61 λόγω μετάφρασης δεν κατανοώ το νόημα της ε, τροπολογίας αυτής. Θεωρώ όμως ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επειδή η έκθεση είναι αρκετά σημαντική και είμαι πεπισμένη ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα αποδεκτό, σαν θετικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, uh, να διευκρινίσω ότι μου είπαν ότι υπό την ενισχυμένη συνεργασία κάθε επιτροπή θα πρέπει να ακολουθήσει αυστηρά το δικό της ε, τομέα πραγματογνωμοσύνης, όπως λέει και ο κανόνας 50 στον ε, κανονισμό του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει δηλαδή να συμφωνήσουμε για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα της κάθε επιτροπής. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποφασίζουν οι πρόεδροι των επιτροπών σε διαβούλευση με τους ηγητές των Γι' αυτό ακριβώς πάρα πολλές από τις ε, τροπολογίες δεν κρίθηκαν αποδεκτές. Η κυρία Μοναστατή. Juste sur ce point, Madame la Πρόεδρε, ευχαριστώ μου δίνετε το λόγο για το γεγονό ότι οι συγητές έχουν γνώση και είναι ενήμεροι για την σφαίρα αρμοδιοτήτων της κάθε επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι παράδοξο η πρόεδρος μας να έχει κάνει αναφορά σε αυτό το θέμα τη στιγμή που στην ίδια συνεδρίαση αποδεχόταν ως ένα θέμα εργασίας για το επόμενο έτος του 2011 την ε, γυναίκες τις λιγότερο γυναίκες που βρίσκονται σε λιγότερο νοική κατάσταση κάτι το οποίο μας αφορά αποκλειστικά για τις γυναίκες δηλαδή. Έχουμε λοιπόν εδώ μια θέση αρχής ενάντια σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες οι οποίες περιλαμβάνουν τον όρο γυναίκα αφενός και αφετέρου στην ίδια συνεδρίαση αποδεχόμαστε ένα θέμα εργασίας πάνω στο οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε του χρόνου για την κατάσταση των γυναικών όσον αφορά την κατάστασή τους ως λιγότερο ευνοημένες στον χώρο εργασίας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια διαφορά θέσης που παρουσιάζει το ίδιο άτομο στην ίδια συνεδρίαση. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Δεύτερον, και από αυτού ήθελα να λάβω το λόγο αμέσως μετά αυτά που είπατε εσείς και γι' αυτό είχα ζητήσει το λόγο. Γενικά λοιπόν, η Πρόεδρος ε, να πω και πάλι ότι έχουμε την ισχυμένη συνεργασία και είχε γίνει η συμφωνία. Θα προσπαθήσω να λάβω διευκρινήσεις από την κυρία Μπερές, την Πρόεδρο, για τα θέματα που έθιξε στην συνάντηση των συντονιστών. Εγώ δυστυχώ έλειπα από τελευταία συνάντηση των συντονιστών, οπότε δεν ξέρω ακριβώ πριν ε, περί τίνο πρόκειται. Θα κοιτάξω πάντω να λάβω διευκρινήσει. Πάντω. όσον αφορά αυτή την έκθεση, έχουμε την ενισχυμένη συνεργασία και συμφωνήθηκε μεταξύ των Προέδρων των δύο Επιτροπών Δικαιωμάτων Γυναικών, πολιτικέ ίσων ευκαιριών συμπεριλαμβανομένε τη μεταξύ άνδρων και γυναικών σε σχέση με, την, με τι ευκαιρίε στην αγορά εργασία και η αντιμετώπιση του στον χώρο εργασία. Αυτή είναι νομίζω η αρμοδιότητα τη Επιτροπή των Γυναικών. Και γι' αυτό ακριβώ αποφασίστηκε από την Επιτροπή Γυναικών και από την πρόεδρο τη Επιτροπή μα να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών. Έχουμε την κυρία, κυρία Μωράν Σατέ. Κυρία Μωράν Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, τον πέρεψα γιατί είχαμε και ένα διαδικαστικό και τέλο πάντων. Ευχαριστώ. Όχι, διαδικαστικό πρώτα. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου που δεν αφορά μόνο το σημερινό συμβάν αλλά γενικότερα πολλές εργασίες της Επιτροπής μας φαίνεται να υπολείπονται των εργασιών άλλων επιτροπών στις οποίες εμείς δεν συμμετέχουμε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί οι αρμοδιότητες Επιτροπής Απασχόλησης που είναι ξεκάθαρες, αγοραργασία κλπ. κλπ γιατί τα έχουν ιδιοποιηθεί αυτά τα θέματα άλλες επιτροπές που ασχολούνται με άλλα θέματα. Τα θέματα που αφορούν αγορά εργασία είναι αρμοδιότητα της δικής μας επιτροπής. Η κοινωνική ένταξη είναι θέμα δική μας επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να λάβω μια πρόσθετη εξήγηση, όχι μόνο για αυτό το συμβάν, αλλά γενικότερα. ενδεχομένω θα πρέπει να κάνουμε μια έτσι γενικότερη σκέψη για αυτά τα θέματα. Και καταλήγω, είναι προφανές ότι το άρθρο 50, το άρθρο 50 λέγω, μιλά για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ διαφορών ε, επιτροπών, όμως πάντοτε στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων. Ναι, μπορώ να συμφωνήσω με αυτό το σημείο για εσάς. Και εγώ αναρωτιόμουν τι συμβαίνει. Θα πρέπει να το θέσουμε όμως στη διάσκεψη των Προέδρων πολιτικέ ομάδε θα πρέπει να το παρουσιάσουν εκεί. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο πριν από τι ψηφοφορίε. Ε, λοιπόν, εάν δεν είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό διαδικαστικό, αλλά θα πάρω το χρόνο αυτό από το χώρο αγορευσή σα, αν ε, μακριούρεστε. Το πρώτο θέμα, πρώτα, είναι ότι ο τρόπος λειτουργίας που, στον οποίο αναφερθήκατε ισχύει για τις ε, εκθέσεις νομοθετικού περιεχομένου. Λοιπόν, δεν έπρεπε επουδενή να υπάρχει όρος γυναίκες στις τροπολογίες. Μου είπαν, δηλαδή δεν μπορεί να φέρει τη γυναίκα σε μια έκθεση για το πρόσωπο για στόχιας. Ε, τρελαθήκαμε θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις τροπολογίες 27, 45 και 54 που α, μη παραδεκτές για αυτό το λόγο, αλλά νομίζω αυτό είναι θέμα ουσιαστικότατο της Επιτροπής Απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξεταστεί το κατά πόσο είναι πραγματικά αποδεκτές ή όχι αυτές οι τροπολογίες. Εξ ονόματος της κυρίας Γκρούνη και της υποφαινομένης θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στην τροπολογία 71 η οποία αναφέρεται σε ένα ελάχιστο εισόδημα παρά μου δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα. Λοιπόν, 71 είναι αυτή η τροπολογία, πρέπει να την προσέξουμε. Δεν συμφωνούμε. Και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπάρχουν οι τροπολογίες 22, 23 και 26 που αναφέρονται στο ότι είμαστε εμείς υπέρ της μείωσης του ταμείου αυτού, πράγμα που είναι απαράδεκτα. γιατί δεν θα ήταν κάτι τέτοιο σύμφωνα με τους στόχους μας κοινωνικής συνοχής. Και θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στην τροπολογία που αναφέρεται στην επικουρικότητα. Όσον αφορά κατά πόσο οι τροπολογίες είναι αποδεκτέ ή όχι, εγώ θα ήθελα πρόεδρε να ζητήσω μια ψηφοφορία για να ξέρω ποιοι συμφωνούν. αυτέ οι τροπολογίες ε, να επιστραφούν στην Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ κύριε Ατόρα. Благодаря, госпожо председател. Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση γι' αυτό γιατί διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκαν αυτά τα θέματα φτώχεια και γυναίκες. Δεν συμφωνώ. Διότι εδώ το θέμα είναι η ανέχεια μεταξύ των γυναικών στην Ένωση. Επομένως εδώ μας αναγκάζουν να χωρίσουμε δύο θέματα που συνδέονται από τη φύση τους. Μας είπαν ότι οι επιτροπές αυτές αποφάσισαν να κατανείμουν τα θέματα όπως είπαμε. Εγώ δεν έχω λάβει τέτοια επιστολή όμως. Η συντονίστριά μας διαμαρτυρήθηκε και νομίζω ότι ένας τέτοιος διαχωρισμός δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Λυπούμε γιατί η κυρία Τσίμερα που ουσιάζει, γιατί μας έχει πει βέβαια ποιες τροπολογίες απορρίπτει, έχει προτείνει συμβιβασμούς, αλλά δεν καταλαβαίνω τη συμφωνία αυτή. Και οι σοσιαλιστές ήταν κατά τις 22, γιατί εδώ πρόκειται για τον προϋπολογισμό από τη μία και από την άλλη λέμε ότι δεν χρειαζόμαστε κανένα κονδύλιο για την καταπολέμηση της ανέχειας των γυναικών. 22, 23 και 25, όχι 26, θα μπορούσαν να συνδυαστούν σε ένα συμβιβασμό που να κανονίζει τις δαπάνες του κοινωνικού ταμείου. Δεν ξέρω τι πιστεύετε λοιπόν συνάδελφοι, εγώ όμως νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε την πρόταση που ακούστηκε πριν από λίγο και πρέπει να ξαναγίνει η συζήτηση. Εγώ διαφωνώ με τη συμφωνία που έγινε. Νομίζω ότι το πρόσωπο της γυναικείας ανέχειας είναι γενικότερα το πρόσωπο της ανεχίας. Υπάρχουν ε, χωρισμένες, υπάρχουν ανήπαντρες μητέρες, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να θίξουμε εδώ και τα περισσότερα αφορούν την Επιτροπή μας. Προσπάθειες να κρατηθούν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, να αντιμετωπίσουν παράλληλα το πρόβλημα της ανατροφής των παιδιών τους, τέτοια πράγματα. Γι' αυτό υπέβαλα σχετικώς τροπολογίες. Όσο για την, τον μη αποδεκτό χαρακτήρα ορισμένων, μερικές τροπολογίες τις ε, κρίναμε πολύ αυστηρά. Ότι δεν μπορούν δηλαδή, δεν μπορεί η Επιτροπή Απασχόληση να μιλήσει για γυναίκες, τι πράγματα είναι αυτά. Φυσικά κοινό στόχος ολοκλήρου του Κοινοβουλίου είναι να γίνει μια όσο πληρέστερη έκθεση γίνεται. Και όταν λένε ότι η Επιτροπή Απασχόλησης φοβάται μήπως υπάρξουν επικαλύψεις, σωστό είναι αυτό. και η Επιτροπή Γυναικών ενδιαφέρεται περισσότερο από κάθε άλλη να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Είμαι και εγώ συντονίστριά της και ξέρω ότι πολλοί στην Επιτροπή μας εδώ είναι μέλη και της Επιτροπής Γυναικών, πολλές μάλλον. Και θα μπορούσα εγώ να δεχτώ πολλές από τις τροπολογίες εδώ και στην Επιτροπή Γυναικών. γιατί πολλές από τις τροπολογίες είναι θετικές ακόμη και του ΕΛΚ και θα το να ψηφιστούν εδώ ή στη γυναικών δεν είναι το πιο ενδιαφέρον, δεν με αφορά. Αν η έκθεση καταλήξει να βελτιωθεί, τίνω να συμφωνώ με όλους σας προσωρινά προεδρεύω, αλλά θα το θέσω στην κυρία Μπερές, εκείνη πήρε την απόφαση και έκανε τη συμφωνία με την πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών και τους εισηγητές να απορριφθούν οι τροπολογίες. Λοιπόν, θα το ξαναθέσω με την πρόεδρο ώστε πριν την ψηφοφορία να τις ξαναδούμε. Γιατί συμφωνώ. Η γραμματεία δεν είναι βέβαιοι ότι είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες και ότι πρέπει να διαχωριστούν τα θέματα τόσο απόλυτα. Θα το ξαναπώ λοιπόν στην κυρία Μπερές ώστε να ξαναδούμε αυτά. Ο κύριος Σέρκης. Δεν ζήτησα το λόγο, αλλά μια και μου το δώσατε να πω ότι συμφωνώ. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που πάμε σε θα πρέπει να ζητήσουμε διευκρινήσει. Ευχαριστώ πολύ η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχή που συμφωνήσατε να τεθεί το θέμα στη συνεδρίαση των συντονιστών και να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί πήραμε όλοι αυτό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και, είμαι, και εγώ μεταξύ εκείνων που εξεπλάγησαν από την αποχώρηση αυτών των τροπολογιών και δεν κατάλαβα γιατί ακριβώς. Ε, γιατί ε, υπήρχε και μια πράσινη τροπολογία που δεν ξέραμε ακριβώς πού θα πρέπει να υποβληθεί ή όχι. Και εγώ είπα ότι εντάξει μπορώ να αποσύρω κάποιες από τις δικές μου τροπολογίες. Αλλά τώρα δεν καταλαβαίνω πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε. Να ξαναστέλνουμε ηλεκτρονικά ταχυδρομείο και να πω εντάξει δεν α, αποσύρω. Αποσύρω την απόσυρση, τι θα πρέπει να κάνουμε, πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατάσταση αυτή. Πρόεδρος, να σας απαντήσω σε αυτό. Όλες οι τροπολογίες θα επανεξεταστούν και θα σας ειδοποιήσουμε το γλυγορότερο δυνατόν κατά πόσον έχει αλλάξει κάτι. Αυτό είναι νομίζω πολύ σωστό, γιατί πολλοί εδώ έθιξαν αυτό το θέμα. Και προφανώ και εγώ έχω την ίδια εντύπωση που έχετε και εσεί, ότι θα πρέπει δηλαδή να εκτάσουμε κάθε μεμονωμένη τροπολογία και να δούμε κατά πόσο αυτέ οι τροπολογίε μπορεί να υποβληθούν στην Επιτροπή Απασχόληση ή όχι και θα σας ειδοποιήσουμε το γλυγορότερο δυνατόν, για να ξέρετε αν άλλαξε τίποτα ή όχι. Ο κύριος Μάν, θα είμαι σύντομο. Γιατί ακριβώς θέλω να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν θέλουμε να είμαστε αναγκασμένοι να εργαζόμαστε τόσο στενά που ο όρος γυναίκες να επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο από την Επιτροπή των γιατί έχουμε παραδείγματο χάρη και την Επιτροπή Πολιτισμού που ανήκει και η νεολαία και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τον όρο νεολαία. Ε, εμείς, παρόλο που η ανεργία, η ανεργία των νέων. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σαν να μέσα στο καρναβάλι. 11 Νοεμβρίου αρχίζει το καρναβάλι στη Γερμανία, αλλά εδώ νομίζω αρχίσαμε ήδη. Λοιπόν, θα πρέπει να υποβληθούν οι τροπολογίε κατά δυνατόν περισσότερε επιτροπέ που ασχολούνται με το θέμα αυτό, ε, με τον κίνδυνο ότι μπορεί κάποια στιγμή να καταψηφθούν. Λοιπόν, αυτά. Ε, παράγραφος 15. Εντάξει, ενδυναμωμένη συνεργασία επίσκερο. Αλλά η κ. Σεράν είπε ότι θέλει να δράσει ένα ε, να εγγραφεί εδώ, αλλά αυτό που θέλουμε εδώ είναι μια γραπτή απάντηση. Το λέω προς την Κομισιόν ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα το πάρετε, λέει η Πρόεδρος. Θα φροντίσουμε. Η κυρία Φιγκερά. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Όπως και η συνάδελφος Κορνέλισεν, είμαι και εγώ συντονίστρια στην Επιτροπή Γυναικών από πολιτική ομάδα και είμαστε μέλη και σε αυτή την Επιτροπή εδώ. Γνωρίζουμε λοιπόν το πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών βεβαίως θα πρέπει να δώσει τη δική της ε, γνωμοδότηση και είναι σημαντικό να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Η Επιτροπή λοιπόν των γυναικών και αυτό είναι και η γνώμη της κυρίας Μπάουερ που αντιμετωπίζει την διακατάσταση, δηλαδή είναι ε, μέλος στην Επιτροπή Γυναικών και συντονίστρα μάλιστα δεν κάνω λάθος. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχουμε πρόθεση να μην αφήσουμε την Επιτροπή Απασχόλησης να κάνει τη δουλειά της. Ιδιαίτερα στον τομέα αυτό που είναι και σημαντικός, γιατί το κυριότερο ζήτημα της νομοδότησης αυτής είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή η φτώχεια των γυναικών. Όμως θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία στην Επιτροπή μας, εδώ στην Επιτροπή δηλαδή Απασχόλησης, για να ακολουθήσουμε αυτή ακριβώς την αρχή. Και γι' αυτό ακριβώς συμφωνώ να περιλάβουμε εδώ τις προτάσεις που οι συνάδελφοι της Επιτροπής Απασχόλησης θα καταθέσουν και που αναφέρονται και αυτές τις προτάσεις στη φτώχεια των γυναικών, εκτός βεβαίως από το κομμάτι που αφορά τη δουλειά που θα κάνει η Επιτροπή Γυναικών. Και στη συνέχεια σε τελική ανάλυση αυτός που είναι αρμόδιος επί της ουσίας θα πρέπει να είναι κάπως λογικός και θα πρέπει να δεχτεί τις διάφορες προτάσεις που θα κατατεθούν ώστε να αποφευθούν οι επικαλύψεις. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν η πιο σωστή απόφαση. Να υπάρχει κάποια λογική δηλαδή, χωρίς να υπάρχει έτσι πόλεμος μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Η Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση είναι κάπως παράξενη. Για αυτά τα θέματα που επικαλύπτονται όσον αφορά την αρμοδιότητα των επιτροπών, παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε την ενισχυμένη συνεργασία και είναι αλήθεια ότι αυτή η συνεργασία δεν ήταν πάντοτε ομαλή. Κυρίως σε περιπτώσεις όπως αυτή που είναι αδύνατον να διαχωρίσουμε τις αρμοδιότητες των δύο επιτροπών. Όμως ποτέ στα έξι χρόνια ποτέ δεν είδα μια παρόμοια πρακτική, δηλαδή μια επιτροπή να αποφασίσει να στείλει στην άλλη επιτροπή πίσω τις τροπολογίες της. Φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση η διαχωριστική γραμμή είναι, πώς να το πω, να το πω, πολύ ευέλικτη και είναι αδύνατο να βρούμε έτσι μια ακριβή διαχωριστική γραμμή. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε περισσότερη καλή θέληση για να λύσουμε το θέμα αυτό και αυτό θα το χρήσιμο αντί να καθόμαστε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Ευχαριστώ. το αυτό το θέμα. Και θα να σας... Α, όχι, συγγνώμη. Κύριε Κόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ξεχάσατε. θα ήθελα να πω δύο λόγια, όχι για τις τροπολογίες, αλλά δεν άκουσα τίποτα για την καταβολόμηση της φτώχειας με τη δημιουργία μιας ισχυρούς ε, οικονομίας. Γιατί η αγορά απασχόλησης βελτιώνεται όταν υπάρχει ισχυρή βιομηχανία. Οι γυναίκες δεν ζουν σε ένα κενό. Για να καταπολεμήσουμε λοιπόν τη φτώχεια των γυναικών και όλων των υπολείπων, πρέπει να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη των ε, θέσεων απασχόλησης και την ε, άθυση της οικονομίας. Λοιπόν, για να καταπολεμήσουμε την φτώχεια, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τα προβλήματα της συγκεκριμένα που υπάρχουν λόγω της φτώχειας, λόγω της ανοιχίας. Και εδώ βέβαια έχουμε το θέμα της ε, Θα ήθελα εγώ να αναφερθώ συγκεκριμένα στην τροπολογία με υπαριθμό 22, που νομίζω αξίζει να, της προσοχής σας, ο λόγος για τον οποίο ε, λέω ότι δεν πρέπει να αυξήσει το κοινωτικό κοινωνικό ταμείο αυτή τη στιγμή, γιατί τα χρήματα αυτά από πού θα προέρθουν από τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να αυξήσουν τους προπολογισμού τους. Και όπως είπα, ότι το καλύτερο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τα κράτη-μέλη στο δικό του επίπεδο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, γιατί αυτά καλύτερα ξέρουν τι γίνεται στι χώρε αυτέ. Και επίση δεν συμφωνώ με αυτόν τον όρο σημαντική αύξηση. Θα ψηφίσουμε δηλαδή να αυξηθεί σημαντικά. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αποχωριζόμαστε από την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε να αυξηθεί κάτι σημαντικό, α πούμε τουλάχιστον Πόσο είναι το σημαντικό αυτό, ποιο ποσό προβλέπουμε. Γιατί έτσι αυτό είναι τελείως ασαφές και είναι πραγματικά σαν να ζου, ζείτε σε διαφορετικό κόσμο από εκείνο στον οποίο ζω εγώ. Επίσης θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία 51 που διαγράφει το σημείο 5. Πάλι, γιατί δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η κοινωνική προστασία και η κοινωνική πολιτική συμβάλλουν στην ελάττωση του βάθους και της διάρκειας της ύφεσης. Κανέ, κανένα, κανένα αποδεικτικό στοιχείο για κάτι τέτοιο και γι' αυτό θα πρέπει νομίζω να διαγραφεί αυτό το σημείο 5. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα εγώ σας ευχαριστώ. Η, η έγκριση στην Επιτροπή απασχόληση θα γίνει σε 9 Νοεμβρίου. Θα πρέπει να συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα το θέμα και θα ήθελα επίση να ζητήσω από όλους να προχωρήσουν και να έρθουν σε επαφή με του επικεφαλεί των πολιτικών ομάδων για να αλλάξει η κατάσταση στα πλαίσια της ε, διάσκεψης των Προέδρων. Γιατί αυτοί έχουν την ευθύνη. Εγώ θα το θίξω το θέμα με την κυρία Μπερές, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσείς να το θίξετε εναντί των επικεφαλής των δικών σα πολιτικών ομάδων. 9 Νοεμβρίου είπαμε. Θα ψηφίσουμε πάνω σε αυτό στην Επιτροπή μας. Back to Mr. Handel. ich kann nur so viel sagen. Εγώ να σας πω ότι παρακολούσα στενά την συζήτηση σημειώσαμε αυτά που είπατε και θα κάνω ό,τι μπορώ για να ενημερώσω την κυρία Τσίμερ για τη συζήτηση εδώ, ούτως ώστε να τα λάβει υπόψη στη δική σας περαιτέρω εργασία. Ευχαριστώ. Right, thank you very much for that. And now we come to the next item. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης θα ψηφίσουμε όλα μαζί τα θέματα όπως έχει συμφωνηθεί από την ομάδα εργασίας και όπως ξέρω δεν υπάρχουν προβλήματα με καμία πολιτική ομάδα. Λοιπόν, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά νομίζω. Παρακαλώ, αν δεν έχετε την κάρτα σας πέστε μου. Και για τις 7 επιστολές, παρακαλώ, έχετε η ψηφοφορία. Uh, Έληξε. Τριάντα τέσσερις υπέρ, δύο κατά. Καμία αποχή. Ευχαριστούμε επόμενο θέμα για να δω που το είχα. Για τα συστήματα συνταξιοδότησης. Η συγγήτρια και η Όμεν Ρόιτεν δεν είναι εδώ. Άρα θα κάνουμε ένα-δυο λεπτά διάλειμμα ώσπου να έρθει. Παρακαλώ λάβετε θέσεις. Έρχεται η κυρία Όμεν Ράιτεν, ήρθε μάλλον. Αρχίζουμε λοιπόν προς μία επαρκή και ένα ασφαλές σύστημα συνταξιοδότης στην Ευρώπη. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Όμεν και Ρόιτεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουμε μία πράσινη βίβλο που βασίζεται σε οδηγία που αυτή τη στιγμή έχει παγώσει στο Συμβούλιο για την κινητικότητα και τους διάφορους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των συντάξεων και τη βιωσιμότητα του συστήματος. Συνεργάστηκα με τη Γραμματεία και με διάφορους εμπειρογνώμονες και την έκθεση θα τη στείλω την επόμενη εβδομάδα στη μετάφραση. Προσπάθησα να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα που τίθενται και η απάντηση μπορεί να μην αποτελεί λύση του τωρινού προβλήματος αλλά θα ανταποκρίνεται στα προβλήματα αυτά και θα προσβλέπει προς το μέλλον. Ελπίζω, Πρόεδρε, όταν η έκθεση τελειώσει, να μπορέσουμε να διαβουλευθούμε και τους κοιόδης των διαφόρων ομάδων για να καταθέσουμε τροπολογίες αν χρειαστεί ώστε να καταλήξουμε σε μία συνεπή άποψη του θέματος. Τι εννοώ. Εγώ ως εισηγήτρια θα προσπαθήσω όλα αυτά να τα θέσω ρητά σαφώς και καθαρά, όχι μόνο συμβιβασμούς και μόνο συμβιβασμούς. Έτσι ώστε να υπάρχει, να δοθεί μια συνεπής απάντηση στο θέμα του μέλλοντος των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που τίθεται είναι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, χρειάζεται να κάνει κάτι για να αλλάξει τα ισχύοντα στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη ιδιαίτερα αν το συγκρίνουμε με το, αυτά που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Διότι εάν τα συνταξιδοτικά συστήματα δεν είναι βιώσιμα, αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, στους προϋπολογισμούς των χωρών μελών. Άρα, χρειάζεται εδώ μια ευρωπαϊκή απάντηση. Αυτό δεν σημαίνει, Πρόεδρε, ότι πρέπει η Ευρώπη να καθορίσει άτεγκτα όλους τους κανόνες αλλά τουλάχιστον πρέπει να δώσει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για το, την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει και θέλουμε να κινηθούμε. Έχουμε μπροστά μας μία ανεστραμμένη πυραμίδα δηλαδή οι νέοι σε αυτό το σύστημα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε pay as you go είναι όλο και λιγότεροι και θα χρειάζεται να χρηματοδοτήσουν παρόλα αυτά όλο και περισσότερους ηλικιωμένους. Έτσι θα υπάρχουν πολύ λιγότερες εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Στις περισσότερες χώρες λοιπόν η ηλικία συνταξιοδότησης είναι χαμηλότερη, η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης είναι χαμηλότερη από την επίσημα προβλεπόμενη. Και αυτό σημαίνει ότι τίθεται το ερώτημα αν πρέπει να τεθεί μια πανενοσιακή ηλικία συνταξιοδότησης. Το προσδόκιμο ζωής όμως διαφέρει από χώρα σε χώρα και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και βιώσιμο σύστημα και όπως λέει και η Κομισιόν πρέπει να είναι και επαρκές. Και εμείς ανέκαθεν λέγαμε 60% του μέσου εισοδήματος να είναι η σύνταξη. Αυτό όμως δεν είναι δεδομένο, διότι θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να καθορίζουν ποιο είναι το επαρκές ποσοστό. Αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να το θέσουμε πανενοσιακά. Επαρκής σύνταξη θα πρέπει να καλύπτει τους τρεις πυλώνες. Λοιπόν, ασφαλές και βιώσιμο συνταξιδοτικό σύστημα. Σε μερικές χώρες μέλη έχουν και τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα, ενώ στις νεότερες χώρες μέλη ο δεύτερος αυτός πυλών δεν είναι πραγματικός δεύτερος πυλών. Και αυτό το έχω δει σε πολλές περιπτώσεις. Λαμβάνονται υπόψη ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας όπου είχε καθορίσει παλαιότερα η Παγκόσμια Τράπεζα για τις χώρες αυτές και οι χώρες αυτές τώρα, τώρα που βασικά εφαρμόζουν το 1α και 1β ως πυλώνες τώρα έχουν πρόβλημα διότι στον πρώτο πυλώνα υπάρχει το σύστημα Pay as you go ενώ στον δεύτερο γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων, αλλά το χάσμα είναι τόσο μεγάλο ώστε αυτά που εξοικονομούνται βγαίνουν από τον προϋπολογισμό και ξαναμπαίνουν στον πρώτο πυλώνα. Αυτό δεν προβλεπόταν αρχικά. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα άλλες χώρες μέλη πάλι όπου ο πρώτος πυλώνας ε, λειτουργεί πολύ καλά και έχουν εξοικονομηθεί εκατοντάδες δισεκατομμυρίων και αυτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον δεύτερο πυλώνα. Γιατί? Διότι το χρηματιστήριο δεν είναι τόσο υγιές όσο προβλεπόταν και δεύτερον διότι μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων ζουν περισσότερο χρόνο. Και αυτό πιέζει, πιέζει πολύ. Γι' αυτό νομίζω πρόεδρε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα, συνεργαστήκαμε με την Επιτροπή Εικόν και πρέπει να δούμε και την οδηγία ΙΟΡΠ που είναι δικαιοδοσία της εικόνος αλλά εδώ υπάρχει ανάγκη να το δούμε και η ασφάλεια, η ασφάλεια των συντάξεων η επιτήρηση των κονδυλίων και ξέρω ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορεί να μην συμφωνούν. Η επιτήρηση των κονδυλίων αυτών είναι κάτι το απαραίτητο μέχρι κάποιο βαθμό. Και γιατί αυτό, διότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι ένα τέτοιο ταμείο είναι απλώς κάτι που επηρεάζεται από την εθνική αγορά, επηρεάζεται και από την ευρωπαϊκή αγορά. Και κάτι άλλο που θέλω να προσέξουμε είναι ότι όταν μιλάμε για συντάξεις, οι νέοι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη σύνταξη ακόμα, γιατί δεν ξέρουν και πολλά περί αυτής. Άρα χρειάζεται και μεγαλύτερη πληροφόρηση. Θα έπρεπε λοιπόν να δώσουμε την ευκαιρία αφού, αφού θα έχουν μιλήσει και οι κοινωνικοί εταίροι να κάνουμε και μεγαλύτερη πληροφόρηση προς τους νέους. Ευχαριστώ. Και τώρα οι κοινωνικοί εταίροι. Η Ρεβέκα Σμίθ από το Business Europe. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή Απασχόληση που μας δώσανε τη δυνατότητα να έρθουμε εδώ και να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας η Business Europe προετοιμάζει αυτή τη στιγμή, τελειοποιεί από την πράσινη βίβλο. Θα σας πούμε πάντως κάποιες από τις ιδέες μας. Καταρχήν, θα να σχολιάσω τρεις τομείς. Καταρχήν την ανάγκη μεταρρύθμισης των συνεξιωτικών ε, συστημάτων στα κράτη-μέλη και επίση ότι εμεί αισθανόμαστε εντονά ότι χρειάζονται περαιτέρω μέτρα από τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλιστεί η εφορία των ε, συστημάτων αυτών και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να μειωθεί το δημόσιο χρέο και να ε, εξασφαλιστεί η εφορία των δημόσιων οικονομικών στο μέλλον. Έχουμε εδώ μια μεταρρύθμιση των αγορών απασχόληση και είναι σαφές ότι αν μεταρρυθμίσουμε τα συνταξιωτικά συστήματα, εμείς θα θέλουμε οι άνθρωποι να εργάζονται περισσότερο, πιο μακρά δηλαδή στη ζωή τους, άρα θα πρέπει να έχουμε από την άλλη μεριά καλές θέσεις απασχόλησης, ε, ανάπτυξη και να υπάρχουν και θέσεις απασχόλησης ιδιαίτερα για τους πιο ηλικιωμένους. Μετά το άλλο ήμιση της Πράσινης Βιβλίου που είναι το θέμα των ε, συντάξεων από τις εταιρείε της ίδιας. Για μας η κύρια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν να ενθαρρύνει τα κρατημένα να λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν την ε, σταθερότητα και εφορία των συναξιωτικών συστημάτων. Αν τα κράτη-μέλη δεν αλλάξουν τις ε, τακτικέ και διατηρήσουν τα επίπεδα στα σημερινά, υπάρχουν τεράστια προβλήματα λόγω και της, ε, του προσδόκιμου ζωή των ε, εργαζομένων. Συμφωνώ με αυτό που είπε η συγχύτρια, ότι δεν πιστεύουμε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ορίσει ποιο είναι το σωστό εισόδημα κατά τη ε, διάρκεια της συνταξιδότησης θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι υποχρεωτικές συντάξεις ε, τα τελευταία χρόνια δίνουν το 70% του μέσου όρου των ανθρώπων, ε, των, ε, του μέσου όρου, συγγνώμη, του τελευταίου μισθού εκείνου που έχουν υψηλά εισοδήματα και 80% εκείνου που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Θα πρέπει να εξακολουθούν να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη, όπως έγινε το τελευταίο μήνες, τα τελευταία χρόνια, σε μια επιγόντως αναγκαία μεταρρύθμιση των δημοσίων οικονομικών η Κομισιόν υπέβαλε κάποιες ε, ε, προσωμιώσεις ε, στο τομέα αυτό και είδε ότι κατά μέσο όρο θα αυξηθεί κατά 4-7% του ΑΕΠ η δαπάνη των κρατών μελών και σε ορισμένες χώρες μάλιστα 7%. Και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε βέβαια τις δικαιώματα λόγω των προβλημάτων αυτών των δημοσίων οικονομικών. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ότι θα πρέπει να εργάζονται μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους οι εργαζόμενοι. Η αύξηση της ε, διάρκειας ε, συναξιοδότηση ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. 20 από 20 έως 25 χρόνια στις γυναίκες και 14 24 στους άντρες από την άλλη μεριά ε, θα μπορούσαν να υπάρχουν χαμηλότερα έσοδα κατά τη διάρκεια της ψηλότερε υψηλότερες ε, συμβολές και συνεισφορές. Αυτές όμως δεν είναι οι πιο κατάλληλες λύσεις κατά τη γνώμη μας. Και το να αυξηθεί η ηλικία συνταξιδότηση στα κράτη-μέλη είναι η πιο κατάλληλη λύση. Και οπωσδήποτε θα πρέπει τα κράτη-μέλη, ελέγχθη αυτό ήδη, αφενός να αυξήσουν την ηλικία συνταξιδότησης, από την άλλη μεριά να υπάρχουν κάποια μέτρα που θα μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να ε, τηρήσουν αυτά τα όρια. Όπω είπα, αναγνωρίζουμε ότι ε, χρειάζονται μέτρα στην αγορά απασχόληση Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10% ανεργία. Και για τη δημιουργότητα της διατήρησης του σύστηματος ε, Pay As You Go θα πρέπει κάτι οπωσδήποτε να αλλάξει λόγω της Θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά αυτή αποτελεσματικά και να είναι αρκετά ευέλικτη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ευελίκτων συστημάτων ε, συναξιοδότησης στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στις συντάξεις μέσω των ε, των εταιριών ή των συντεχνιών, όχι των κρατικών συντάξεων δηλαδή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μην δεχνάμε ότι υπάρχουν προβλήματα ε, για εκείνους που διακινούνται διαμεθορικά για να εργαστούν και εκεί δεν έχουμε πάρα πολλούς, αλλά τα προβλήματα όσο πάει και παρουσιάζονται πιο έντονα. Η Κομισιόν εδώ, το άκουσα με διάφορες φορές, εξετάζει ήδη κάτι μας στα πλαίσια μιας γιατί ε, μέχρι στιγμή δεν έχει ε, δοθεί απάντηση στην Πράσινη Βιβλία. Θα πρέπει να περιμένει η Κομισιόν νομίζω να δοθούν οι απαντήσει αυτέ, να δει ποια θα είναι η στάση και να δει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Όσον αφορά την κινητικότητα, βέβαια συμφωνούμε όσον αφορά τη σημασία τη αύξηση κινητικότητας στην αγορά εργασία και θα πρέπει να έτσι να ανταποκριθούμε και στην παγκοσμιοποίηση. Η αγορά ε, απασχόληση βέβαια θα πρέπει να είναι πιο δυναμικές η εμπειρία μας ε, δείχνει ότι το θέμα των μελλοντικών συντάξεων είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά εκείνους που ήδη παρουσιάζουν μια κινητικότητα ή που σκέφτονται να μετακινηθούν στο μέλλον. Θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα της βελτίωσης κινητικότητας μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις συντάξεις αυτές από τις διάφορες επιχειρήσεις και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σχέδια εδώ είναι πάρα πολύ φιλόδοξα γιατί κάθε κράτος μέλος έχει δικό της σύστημα. Παρ' αυτά θα μπορούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καταγράψουμε πού κινούνται αυτοί οι εργαζόμενοι. Αυτό προβλέπει βέβαια σημαντική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχει επίση μια πρόταση που προέρχεται από την έκθεση Μόντι όσον αφορά το 28ο καθεστώς ε, των συντάξεων αυτών, των επαγγελματικών αυτών συντάξεων και 27 ισχύοντα συστήματα επαγγελματικών συντάξεων θα υποσκαφθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί το θέμα κατά πόσον υπάρχει ε, ανάγκη ενός κοινωτικού συστήματος και πώς θα λειτουργήσει. Βέβαια, οι εργοδότες ε, θέλουν να δίνουν τις κατάλληλες επαγγελματικές συντάξεις στους ε, παλιούς αλλά και στους μελλοντικούς τους εργαζόμενους. Πολλές φορές αυτές οι συντάξεις είναι τμήμα ενός, ε, μιας δέσμης μέτρων υπέρ του εργαζομένου γενικά. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη ενός συστήματος με πολλαπλούς πυλώνες θα πρέπει να εξεταστεί θετικά. Πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν για τα δεξιωτικά συστήματα, αλλά με το να διαφοροποιηθούν οι πηγές του εισοδήματος τη διάρκεια της αναξιοδότησης είναι νομίζω κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ την οικονομία. Υπάρχει κάποια διχοτομία μέσα στο, στην πράσινη βίβλο, γιατί τονίζουν νέοι κανόνες για την ε, χρηματοδότηση των διαφόρων προγραμμάτων ε, συνταξιδότηση, ιδίω επαγγελματική συνταξιδότηση. Εμείς πιστεύουμε ότι η, βέβαια η, λόγω της ψηλής ανεργίας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα συστήματα pay as you go. Δεν θέλω να μπω στι λεπτομέρειε γιατί προφανώ δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Μα δώσατε μόνο 7 λεπτά, Πρόεδρε. Αλλά η Κομισιόν προτείνει διάφορου τομεί για περιττέρω διακανονισμό των επαγγελματικών ε, συντάξεων, ε, παραδείγματο χάρη συμπληρωματικού ε, κανόνε όσον αφορά τη ρευστότητα. Δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται γιατί πιστεύουμε ότι η... τα ταμεία αυτά στην εξαρτησία λειτουργούν πολύ διαφορετικά από τι ε, ασφαλιστικέ εταιρείε για τι οποίε υπάρχει αυτό ο κανόνα τη ρευστότητα και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναμίξουμε τα μέρη με τα δε. θα... Αν θέλετε να πω σε λεπτομέρειε, θα πω αργότερα. Και μια τελευταία παρατηρήση σε ένα τομέα στο οποίο μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, το θέμα τη χωρίς πληροφοριών και γενικά τη ενημέρωση. Γιατί λόγω της έλλειψης γνώσεων και ενημέρωσης τα κράτη-μέλη μέχρι στιγμή δεν ενημερώνουν του πολίτε όσον αφορά τα εξωτικά συστήματα και τι επιλογέ που έχουν μέσα στα πλαίσια των συστημάτων αυτών και ποιε είναι οι προσδοκίε του για το εισόδημα κατά τη διάρκεια τη σύνταξη. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο λόγω των διαφορών των συνταξιδοτικών συστημάτων, αλλά πιστεύουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, μια υποχρέωση να ενημερώσει τους πολίτε όσον αφορά τα διάφορα εξωτερικά συστήματα, πληροφορίες που θα πρέπει να δοθούν με απλό τρόπο, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξηγήσουν την ανάγκη για μεταρρυθμιστικά μέτρα, στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και αν έχετε ερωτήσεις, ευχαριστώ θα σα απαντήσω σε αυτές. Uh, ευχαριστώ πολύ. Ο από το ETUC, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Νόσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να παρουσιάσουν την άποψή τους και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων που εκπροσωπώ εδώ. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε τεχνικές λεπτομέρειες ως απάντηση στα τεχνικά ερωτήματα που τέθηκαν, αλλά θα ήθελα να αναφέρω αντίθετα κάποιες παρατηρήσεις και να διευκρινίσω ότι αυτό που θα πω σήμερα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων, από την Εκκληστική Επιτροπή που είναι το εκκληστικό μας όργανο και που υιοθέτησε τις απόψεις που θα παρουσιάσω σήμερα και που ήδη έχει διαβιβάσει το ψήφισμά μας στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν, αν θέλετε να τα δείτε γραπτός. Το πρώτο θέμα για το οποίο θα ήθελα να επιμείνω εξ ονόματος των συνδικαλιστικών νόσων αφορά τη συζήτηση για το δημογραφικό θέμα. Βεβαίως υπάρχει η γύρανση ευτυχής συχνά του πληθυσμού. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι καινούριο, το ξέραμε αυτό. Και αντίθετα σε αυτά που πιστεύουμε, οι χώρε μέλη δεν περιμένουν τελευταία στιγμή για να ξεκινήσουν την αναθεώρηση των συνταξιωτικών συστημάτων. Υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις που έγιναν βαθμιαία σε όλες τις χώρες. Αυτή όμως η γύρανση του πληθυσμού δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται, να υπερτονίζεται. Θα πρέπει κυρίως να λάβουμε υπόψη μας μία άλλη σχέση η οποία είναι ουσιώδης για τα σταξιδιώτικά μας ε, συστήματα, ιδιαίτερα για το σύστημα κατανομής, δηλαδή η σχέση της οικονομικής εξάρτησης. Με άλλα λόγια, το πόσοι άντρες και γυναίκες και νέοι και λιγότερο νέοι εργάζονται, ποια είναι η ποιότητα της εργασίας τους και ποια είναι η ποιότητα των αμοιβών τους ή τη χρηματοδότηση των συνταξιδοτικών πραγμάτων και ιδιαίτερα των συνταξιδοτικών ταμείων σε μεγάλο βαθμό εξασφαλίζεται από την εργασία και τα εισοδήματα αυτής της εργασίας. Εξού και η προτεραιότητα που δίνουμε εμείς στη συζήτηση αυτή όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας και την ποιότητα των αμοιβών, των μισθών, γιατί αποτελούν την καθοριστική κινητήρια δύναμη. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να πούμε ότι θεσπίζεται νομοθετικά η εργασία, ότι πρέπει κανείς να δουλεύει πιο πολύ και για περισσότερο χρονικό διάστημα, οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε μια διπλή ευθύνη. Την ευθύνη δηλαδή των εργοδοτών βεβαίως, επειδή η εργασία είναι και δική τους ευθύνη, αλλά έχουμε και την ευθύνη των χωρών μελών όσον αφορά δηλαδή τις πολιτικές τους ανάπτυξης και χωροταξίας που εφαρμόζουν κατά πόσο θα έχετε μέσα μεταφοράς, κατά πόσο θα έχετε κατοικία, εκπαίδευση, παιδεία κτλ. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την εργασία και την πρόσβαση στην εργασία. Για μας λοιπόν το πρόβλημα που σχετίζεται με όλα αυτά δεν δεν είναι και τόσο η αύξηση του ορίου ε, συνταξιδότησης, γιατί σήμερα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάνουμε μία μεταφορά των συστημάτων συνταξιδότησης στα συστήματα ανεργίας. Αυτό όμω είναι άσκοπο. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να βάζουμε κι άλλους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νέους, σε καθεστώς ανεργίας και αυτό είχε αναφερθεί στην διάσκεψη της, της Βαρκελόνης πριν από 10 χρόνια και είναι πάντοτε επίκαιρο ότι θα πρέπει να συμπίπτουν η πραγματική ηλικία διακοπής της ε, δραστηριότητας της εργατικής με την ηλικία, την πραγματική, την νόμιμη ηλικία στις ταξιδοτήσεις. Κάνοντας βεβαίως αυτό το πέρασμα στη συνέχεια και είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό αυτό. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι το θέμα της νομοθεσίας και των νέων νομοθετημάτων. Είναι σαφές για μας, για την Ένωση της Νομοσπονδίας των Δικαλιστικών Ενώσεων, η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης στα νομικά καθεστώτα κοινωνικής πρόνοιας και κυρίως στα συνταξιοδοτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ηλικία συνταξιοδότησης. Δεν μπορούν να πούν δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πώ θα διοργανώσουν τα συνταξιωτικά συστήματα και πώς θα χρηματοδοτήσουν οι χώρες μέλη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως στα πλαίσια του επαγγελματικού συστήματος συνταξιοδοτήσεων, στα ιδιωτικά δηλαδή συστήματα συνταξιοδότησης, η Κομισιόν, α, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αρμοδιότητες και το έχει επιδείξει επανειλημμένως ιδιαίτερα την πρώτη φορά όταν είχαμε την οδηγία 9749 σε σχέση με τη διασφάλιση των συμπληρωματικών συμπληρωματικών μάλλον συντάξεων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους αυτή η οδηγία καθορίζει πραγματικά την διατήρηση της αρχής δεν μιλάει όμως για αξιοποίηση αυτών των συμπληρωματικών δικαιωμάτων. Οπότε εμείς στην Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων είμαστε υπέρ μιας βελτίωσης αυτής της ε, οδηγίας. Έγινε ένα πρώτο βήμα, πολύ ωραία, δεν αρκεί όμως αυτό. Επίσης, η οδηγία που αφορά 2008-94 που μιλάει για τα συμπληρωματικά δικαιώματα των μισθωτών σε περίπτωση που υπάρχει αφαιρεγγιότητα εκ μέρου του εργοδότη και εκεί, και εκεί αυτή η οδηγία καθορίζει μία αρχή η οποία όμως δεν περιλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. μόνο το 30% των δικαιωμάτων διασφαλίζονται. Οπότε και εκεί θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και ήδη το έχουμε ζητήσει αυτό. Για τα υπόλοιπα συμφωνώ με το Business Europe όσον αφορά την οδηγία για την επιτήρηση των ιδιωτικών συνταξιωτικών προγραμμάτων. Θα πρέπει να αποτιμήσουμε τον αντίκτυπο της εφαρμογής αυτής της οδηγίας για να δούμε αν περαιτέρω θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Τρίτο σημείο που θα ήθελα να θίξω εντάχει αν επιτρέπετε αφορά την εξέλιξη των ιδιωτικών συνταξιδιωτικών συστημάτων. Στην πράσινη βίβλο εμφανίζεται ως αναπόφευκτο γεγονός, ως κάτι το μοιραίο, η, η μείωση των, ε, των συντάξεων. Εγώ δεν είμαι μάντης. Πάντως αυτό είναι αρνητικό όσον αφορά τα συμπληρωματικά συνταξιδικά συστήματα γιατί θα περάσουμε από ένα σύστημα οριστικού στρατιωτικού προγράμματος όπου θα διασφαλίζει τη συμμετοχή του ο, ο εργοδότης σε άλλα συστήματα συνταξιωτικά που θα έχουν προσωπικό χαρακτήρα όσον αφορά δηλαδή την συσφορά των εργαζομένων οπότε περνάμε από μια συλλογική ευθύνη σε μια ευθύνη προσωπική, ατομική και Μπαίνουμε εδώ ξεκάθαρα στις χρηματοοικονομικές αγορές με όλους τους κινδύνους που επιφέρει αυτό. Και πράγματι, αν γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος και το βλέπουμε, υπάρχει ένας κίνδυνος για το ύψος των μελλοντικών συντάξεων. Όσον αφορά λοιπόν τη φερικιότητα αυτού του καθεστώτος, συμφωνώ για μια φορά με το Business Europe, και συμφωνώ για το ότι οι κανόνες φερικιότητας που έχουν εφαρμοστεί στα συστήματα ασφάλειας για τους μικρούς ε, κινδύνους δεν είναι κατάλληλα όσο θα έπρεπε να είναι δηλαδή τα συντοξικά συστήματα που αφορούν μεγάλες χρονικές περιόδους. Οπότε και πάλι θα πρέπει να προβλέψουμε κάποια μέτρα, κάποιες δικλείδες ασφαλείας και θα πρέπει να εφαρμόσουμε κανόνες που δεν θα έπρεπε να επιβαρύνουν σημαντικά τις εισφορές και που θα έθεταν ένα φιβάλο ολόκληρο το σύστημα. Πρόεδρε, μακρηγόρησα, αλλά θα ήθελα να συνοψίσω την ομιλία μου και να την επικεντρώσω σε αυτό το κύριο ζήτημα, το οποίο είναι ουσιώδες για μας, δηλαδή στο ζήτημα της ποιότητας της εργασίας. Όχι μόνο την, ε, ε, την απασχόληση των ηλικιωμένων, όπως ακούσαμε, αλλά και την απασχόληση, την εργασία των νέων. Γιατί για να είμαστε παραγωγικοί, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σοβαρά αυτό. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάτι το παράδοξο. Δηλαδή, εισέρχονται εργαζόμενοι αργότερα στην, σε, ηλικιακά στην αγορά εργασία και βγαίνουν νωρίτερα. Και Έχουμε ένα ρητό ε, στα γαλλικά «Κάλιο γαδιδρόδενε παρά γαδιδρογύρευε». Αυτά, Πρόεδρε, είχα να σας πω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας κατευχαριστώ. Βερζίνσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, Βόλοζίνσκι μάλλον. Βρισκόμαστε στη φάση όπου τελειώνουμε πια την ανάλυση μας και θα διαπιστώσετε ότι έχουμε πολλά κοινά με τους προηγούμενους δύο ομιλητές από το Business Europe και την Ευρωπαϊκή Νομοσπονδία Συνδικάτων. Θεωρούμε ότι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση όχι μόνο εθνικά αλλά και ενωσιακά διότι <clears throat> υπάρχει κρίση αλλά και οι δημογραφικές προκλήσεις και πρέπει να υπάρξει κάποια μεγαλύτερη ασφάλεια των συντάξεων. Θα περιοριστώ στα κύρια σημεία της πρασίνης φίβλου. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι, έτσι ως εισαγωγή, ότι πρέπει οι συντάξεις να παραμείνουν δικαιοδοσία των χωρών μελών, να γίνει εδώ σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας ακόμη και αν θεωρούμε ότι υπάρχει ρόλος εδώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο ως καθοδήγηση και συντονισμό. Ιδιαίτερα το θέμα της επαρκούς σύνταξης και της σύνδεσής της με το εισόδημα. Εδώ βλέπουμε ένα ρόλο κλειδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν είναι δικό της καθήκον να καθορίσει ακριβώς σε πανενωσιακό επίπεδο ποιο θα είναι ακριβώς ποια το ποσοστό της σύνταξης σε σύνδεση με το εισόδημα. Πρέπει αυτό να παραμείνει στις χώρες μέλη να αποφασίσουν εάν και πώς θα ακολουθήσουν προσέγγιση πολυπυλωνική. Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και η σύνδεσή της με την γενικότερη κοινωνική διάσταση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο λόγω της φυσική σύνδεση που υπάρχει μεταξύ επάρκειας και αηφορίας των συντάξεων. Το ένα συνδέεται με το άλλο καθώς και με τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών γενικότερα. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, μπορεί να παίξει ένα κεντρικό ρόλο εδώ και υποστηρίζουμε την ε, έννοια της οικονομικής governance. Υπάρχει ανάγκη να εργαζόμαστε περισσότερο χρόνο, αυτό είναι αναπόφευκτο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης, διότι το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι βγαίνουν στη σύνταξη πριν από την επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης. Άρα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας για να είναι αυτές πιο ευέλικτες και να πάψουν πια να υπάρχουν οι πρόορες συνταξιοδοτήσει. Γι' αυτό βέβαια πρέπει να δοθούν και τα κίνητρα στις εταιρείες και τους εργαζόμενους για να παραμένουν στην αγορά εργασίας. Ο προσαρμοστικός μηχανισμός είναι το πρόβλημα. Εδώ πάλι θα λέγαμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της επικουρικότητας και η Ένωση μόνο μία απλή κατεύθυνση να δίνει. Δεν βλέπουμε καμία ανάγκη να αναθεωρηθεί η ισχύουσα οδηγία, αρκεί να γίνει μια καλύτερη αξιολόγησή της για να δούμε αν έχει ελλείψεις και μόνον τότε να δούμε αν χρειάζονται νέοι στόχοι για την κινητικότητα και μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων είμαστε υπέρ της διευκόλυνσης της κινητικότητας της εργασίας στην Ευρώπη γενικότερα. Αλλά θεωρούμε ότι η μεταφορά δικαιωμάτων από χώρα σε χώρα όπως προτείνει η οδηγία δεν είναι σωστή πρόταση. Πρέπει να λυθεί πρώτα το πρόβλημα των δημοσιονομικών φραγμών που υπάρχουν Όσο για την πτώχευση των σπονσόρων, αυτό νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα πανενωσιακού επίπεδου. Και τέλος, πληροφόρηση και συντονισμός, πληροφόρηση των ενδιαφερομένων. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να αναθεωρηθούν τα κριτήρια που υπάρχουν για την ελάχιστη απαραίτητη πληροφόρηση αλλά το βελτιωθεί η ποιότητά των και ιδιαίτερα να χρησιμοποιείται εύληπτη γλώσσα γιατί δεν συμβαίνει αυτό σήμερα. Όποτε έχουμε πληροφορίες δεν είναι σε ευνόητη γλώσσα. Ε, κατ' εμάς η επικορικότητα πρέπει να είναι η αρχή για όλα τα μέτρα που αφορούν τις συντάξεις, αλλά η δυνατότητα κάποιου συντονισμού θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, ιδιαίτερα αν βασίζεται στην εμπειρία που έχουμε ήδη μαζέψει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να λύσω τυχόν απορίες. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο Κάρλος Περέτη από το Eurocard. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Στα πλαίσια της ε, δική μου ένωση έχω να σα πω ότι εμεί συμμεριζόμαστε τον στόχο της Κομισιόν και γενικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για διατηρητέ και ασφαλή συστήματα συνταξιοδότηση. Και επίσης η ιδέα του, της, υπέρ της ιδέας να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ταξιδότηση αυτή, παρόλο που οι εθνικές καταστάσεις ε, κάστοτε είναι πολύ πολύπλοκες. Και γι' αυτό βέβαια η ιδέα του πλαισίου δείχνεται κάπως δύσκολη. Ε, για να προχωρήσουμε προς ένα πλαίσιο θα μπορούσε να υπάρξει καταρχήν η οθέτηση μιας μεθόδου μέσα στα πλαίσια με συμφιλίωσης μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Συμβουλίου. Βέβαια, παρόλο τις κοινωτικές προσπάθειες, το πρόβλημα της απασχόλησης ενός εργαζομένου μεταξύ 55 και 64 ετών είναι πάντα πολύ δύσκολο. Προτού φτάσει κανένας δηλαδή καν στην ηλικία της εγκληματοδόχτησης υπάρχει το πρόβλημα και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε για να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την διάρκεια σταδιοδρομίας. Η κατάσταση είναι η ίδια για όλους. Και για το διοικητικό προσωπικό δηλαδή των επιχειρήσεων, γιατί πολλές φορές οι πιο ηλικιωμένοι μάνατζερ έχουν περισσότερα, ε, περισσότερες ικανότητες κοστίζουν δηλαδή περισσότερο στην επιχείρηση και γι' αυτό καμιά φορά οι εργοδότες προσπαθούν να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους. Εγώ θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι υπάρχει ένα ειδικό πρόβλημα της ισορροπίας μεταξύ των φύλων. υπάρχει μια τομή, αν θέλετε, στις σταδιοδρομίες των γυναικών στην ηλικία αυτή, μεταξύ 55 και 64. Το θέμα που τίθεται λοιπόν είναι πώς θα εμπλακούν όλοι οι τομείς που μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος. Πριν φτάσουν οι εργαζόμενοι στην ηλικία συνταξιοδότησης. Γι' αυτό θα έχουμε κάποιες προτάσεις όσον αφορά το πρόβλημα αυτό στην ε, αγορά, στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν μπορεί να αποφασίσει αντί τα κράτη-μέλη, αλλά δεν μπορεί καν να αποφασίσει χωρίς τριμερή διαπραγμάτευση. Η θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα στρατιωτικά συστήματα θα πρέπει να προβλέπει κάποια στοιχεία κοινωνικής ισορροπίας. Και εδώ ίσως θα μπορεί να αναμειχθεί το ευρωπαϊκό επίπεδο και το εθνικό επίπεδο για τα μέτρα αυτά. Λοιπόν, διαπραγματεύσει στην αγορά εργασία. Και όλα τα άλλα τα ε, σχετικά προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη διαβίου μάθηση Ευρώπη 2020 και ούτω καθεξής. είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξτάσετε το θέμα του χρόνου εργασίας, ούτω ώστε προς το τέλος της επαγγελματικής ζωής να μειωθεί ο, ο ημερήσιος χρόνος εργασίας. Θα ήταν ίσως και αυτό μία λύση για να βελτιωθεί η μετάβαση των εργαζομένων στη συνταξιοδότηση. Κάτι άλλο, αυτά τα λέμε βέβαια σε λεπτομέρειες στο έγγραφό μας. Αλλά δύο συγκεκριμένα θέματα θα ήθελα να θίξω. Είπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποφάσει αντί των κρατών μελών. Από τη μεριά θα μπορούσε και θα έπρεπε να καταστήσει δυνατή την δυνατότητα μεταφοράς αφορολόγητα των συντάξεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κινητικότητα μέσα στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κινητικότητα του επαγγελματικού διοικητικού προσωπικού. Μάνατζερ δηλαδή. Επίσης θα διευκολύνει Ε, την ε, δυνατότητα διευκρινήσεων μεταξύ των Ευρωπαίων και μη Ευρωπαίων εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Ο τελευταίο είναι ο Άντρε Σούμαν, από τους Ευρωπαίους Μάνατζερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσουμε εδώ την απόψή μας. Αρχίζω με μία εισαγωγούλα για την κατάσταση των διαχειριστών των μάνατζερ και των συντάξεών τους για αυτούς. Αυτοί εξαρτώνται πάρα πολύ από τα συστήματα ιδιωτικής συνταξιοδότης για να μπορέσουν να συμπληρώσουν την ανεπαρκέστατη σύνταξή τους. Για να καταλήξουν σε αυτόν τον στόχο ο Ευρωπαίος νομοθέτης μπορεί να συμβάλλει με διάφορους τρόπους. Καταρχήν, το CEC, e η οργάνωσή μας, είναι υπέρ του συντονισμού των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με βάση γενικά πολιτικά κριτήρια όπως την επάρκεια ή βιωσιμότητα, τα γνωστά κριτήρια δηλαδή που υπάρχουν εδώ και χρόνια από την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Επίσης, είχαμε ταχθεί υπέρ της προσθήκης των δύο αυτών στόχων με την ιδέα της ασφαλείας γιατί φοβόμαστε ότι ένα κριτήριο που μπορεί να διαχωρίσει τις ιδιωτικές συντάξεις από τις κρατικές είναι ότι ο εργαζόμενος δεν θα φέρει όλο το βάρος της χρηματοδότησης. Όσο για τη μετάφραση όλων αυτών στην πράξη, της επάρκειας στην πράξη, συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι, δηλαδή ότι τι ακριβώς πρέπει να είναι μια επαρκή σύνταξη είναι θέμα που πρέπει να αφαιθεί στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί οι επαρκείς συντάξεις δεν μπορούν παρά να προκύψουν από το συνδυασμό όλων των πυλώνων και όχι μόνο από συστήματα του πρώτου. Η Ένωση επίσης μπορεί να συμβάλλει θετικά στον τομέα των δημοσιονομικών κανονισμών και στον καθορισμό κοινών κριτηρίων, αλλά εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα διαφορετικά, διαφορετικά συστήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα ένα-ένα εφόσον οι ιδιωτικές και οι κρατικές συντάξεις δεν εμπεριέχουν τους ίδιους οικονομικούς κινδύνους. Οποιαδήποτε εναρμόνιση που θα ξεπερνούσε αυτά που σας είπα, για από τη δική μας άποψη είναι, δεν είναι ούτε απαραίτητη, ούτε επιθυμητή. Αντίθετα, εμείς ελπίζουμε ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στις, στα συντοξιδοτικά συστήματα πρέπει να βασίζεται σε δύο στοιχεία. Πρώτον, θα θέλαμε να υπάρξει κάποιος σεβασμός του γεγονότο ότι υπάρχει πολύ, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στα συστήματα. Και αυτό προκύπτει και από το δικαίωμα που έχουν τα κράτη-μέλη να καθορίσουν τα ίδια τις συντάξεις. Αυτό το λέει και η Πράσινη Βίβλος και το δεχόμαστε και εμείς. Είναι μια αποσαφήνιση χρήσιμη. Δεύτερον, ελπίζουμε επίσης ο Ευρωπαίος νομοθέτης να λάβει υπόψη του τις διαφορές μεταξύ των συνταξιοδοτικών συστημάτων και κυρίως μεταξύ ιδιωτικών και μη. Αυτά δεν είναι θεωρητικά. Και, τα δύο, και οι δύο αυτοί πυλώνες έχουν διαφορές και ομοιότητες και γι' αυτό η εναρμόνιση δεν πρέπει να στοχεύει μακροπρόθεσμα στη συγχώνευση του πρώτου και του τρίτου πυλώνος διότι αυτό θα έβλαπτε δεν θα εξυπηρετούσε τους στόχους ασφάλειας των συστημάτων. Αυτό θα ήθελα να το αποσαφηνίσω τώρα. Με δύο παραδείγματα που τα βλέπουμε συχνά ως προς την πρόσβαση στα δικαιώματα συνταξιοδότης και τη μεταφορά τους. Είναι θεμητό αν θέλει η Ένωση να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να μειώσουν παράλογα υψηλούς φραγμούς. Δεν μπορούν όμως να μειωθούν ή να καταργηθούν χωρίς να ζημιωθούν τα συστήματα κρατικών ασφαλίσεων. Τέλος, η δημοσιονομική επίβλεψη και ο κίνδυνος πτώχευσης. Εδώ αναμένουμε η Ένωση να προσέξει ιδιαίτερα ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι και των δύο συστημάτων συνταξιοδοτήσεων και τέλος να βρει ευέλικτες απαντήσεις, όχι ομοιόμορφες και για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά και τώρα θα επανέλθουμε αφού κάνουν τα σχόλιά τους οι βουλευτές. Πρώτα ο κύριος Σάρκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους φίλους μας που ήρθαν να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους σε αυτήν την τόσο σημαντική συζήτηση. Να αναφέρω δύο σκέψεις ως άτομο που ασχολείται πολλά χρόνια με αυτά τα θέματα στην χώρα μου και παρακολουθώντας ως μάρτυρας αυτά που συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ποιο είναι ο ρόλο της ε, Ευρώπη Αυτά είπε η συγγήτριά μας στην αρχή. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι είναι ουσιώδη ο ρόλο τη Ευρώπη στο θέμα αυτό, παρόλο που ταυτόχρονα θεωρώ ότι λείπουν από την Ευρώπη τα απαραίτητα εργαλεία ώστε η συζήτηση αυτή να φτάσει σε επίπεδο ευθύνη που χρειάζεται. Στην Ευρώπη λοιπόν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο η συζήτηση αυτή να αποδειχθεί επιτυχή στις 27 χώρες μέλη η Ευρώπη θα μπορούσε να συμβάλλει με μια σημαντική προστιθέμενη αξία και να δώσει κάποια έτσι νυφαλιότητα στη συζήτηση αυτή, γιατί στην ε, χώρα μου γίνονται έντονες πολιτικές συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Η Ευρώπη θα μπορούσε να διευρύνει τον ορίζοντα και την προοπτική μας μακροπρόθεσμα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα με τις εκλογές, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις επόμενες γενιές. Θα μπορούσε να προκαλέσει μια πιο νυφάλια συζήτηση η Ευρώπη για τα άτομα τα οποία προσεγγίζουν το θέμα αυτό σε διάφορες χώρες όπου υπάρχει τρόμος από τις συγκυριακές δυσχέρειες. Θα μπορούσε η Ευρώπη να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες, ώστε να μην είναι μόνο σε αυτές τις χώρες όταν θα αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Η Ευρώπη λοιπόν θα μπορούσε να συμβάλλει με μια εκλογήκευση, γιατί έχουμε μια πλούσια ιστορία στην Ευρώπη στα συστήματα συνταξιδότησης. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω αρχικά το εξή. Να προσέχουμε όταν μιλάμε για το θέμα των συντάξεων, ξεχνάμε τα προβλήματα που θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν συντάξεις στην Ήπειρό μα ή τα προβλήματα που θα υπάρξουν στην Ήπειρό αν καταστρέψουμε τα συνταξιοδοτικά συστήματα ή αν τα εξασθενήσουμε. Οι συντάξεις δημιουργήθηκαν επειδή υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Οι δημόσιες συντάξεις δεν είχαν γίνει έτσι στην τύχη. Έγιναν, δημιουργήθηκαν επειδή υπήρχαν εκατομμύρια εκατομμυρίων ηλικιωμένων, ασθενών, ατόμων με αναπηρίες που χωρίς την υποστήριξη αλληλέγγυων συστημάτων πέθαιναν στη φτώχεια. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν αυτά τα δημοτικά συστήματα θα επιστρέψουμε στα προβλήματα που προϋπήρχαν πριν από τη δημιουργία των συντάξεων. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ανυφάλια συζήτηση γνωρίζοντας ότι έχουμε μπροστά μας ένα ουσιώδες εργαλείο για την Ευρώπη οι Ευρωπαϊκέ συνθήκε, Όχι μόνο επειδή, όπως έλεγε η Ρία, επειδή εδώ διακυβεύονται οι προπολογισμοί που είναι σημαντικό θέμα ή επειδή διακυβεύεται η βιωσιμότητα ή τα νομίσματα των χωρών. Εδώ διακυβεύεται ολόκληρη η κοινωνία μας και η επιβίωσή της, γιατί μια κοινωνία που δεν σέβεται τους ορφανούς, τις χείρες, τα δύναμα μέλη της, δεν είναι μια αξιοπρεπής κοινωνία. Και εδώ ακριβώς έχουμε αυτό το πολιτικό στοιχείο. το σύστημα των συντάξεων παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την προστασία των πολιτών. Να μιλήσουμε βεβαίω για την οικονομία, σημαντική η μεταρρύθμιση, να μην ξεχνάμε όμω τι βάσει τη κοινωνική δικαιοσύνη και τη ε, πρόνοια, τη προστασία των πολιτών που είναι η βάση του συστήματό μα. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να κάνουμε μια προσέγγιση λίγο πιο αυστηρή σε αυτό το θέμα. Δεν ε, θέλουμε να πάρουμε το σκάλπ εδώ. Μάλλον, συγγνώμη, δεν, θα, θέλουμε να, να σφάξουμε τον ασθενή εδώ με πολύ δυνατές και ισχυρές λύσεις. Και τέλος Πρόεδρε, να πω το εξή. Αντιδρούμε όταν μιλάμε για τα θέματα τα δημογραφικά, επειδή θα αφιερώσουμε περισσότερα κονδύλια στις συνταξιοδοτήσεις και στις συντάξεις. Γιατί όχι, αν θα έχουμε διπλάσιο αριθμό ηλικιωμένων τα επόμενα 50 χρόνια, θα πρέπει να δώσουμε τα διπλάσια χρήματα. Αν η Ευρώπη θα είναι γυρεότερη, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε αυτή την γυρασμένη κοινωνία. Διαφορετικά θα καταδικάσουμε τους ηλικιωμένους σε 50 χρόνια να ζούσουν με λιγότερους πόρους. Αν λοιπόν η Ευρώπη γερνάει, τότε θα πρέπει να αντιδράμε στο γεγονός ότι θα πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα. Θα πρέπει να προβλέψουμε νέα έσοδα για αυτές τις νέες κοινωνικές ανάγκες. Δεν γίνεται λοιπόν αν το καράβι είναι γεμάτο από ευθύνε, τότε θα μπορούσαμε να σώσουμε το καράβι ρίχνοντα στη θάλασσα τα δύναμα, τα δύναμα μέλη τη κοινωνία, του ηλικιωμένου, χείρε, ορφανά κλπ. Θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή εδώ. Βεβαίω, να κάνουμε περικοπέ. Αλλά γιατί να μην αφιερώσουμε την, τη μισή μα προσπάθεια στην βελτίωση των πόρων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να συμβάλλει με μια λογική και μια ανυφολιότητα στη συζήτηση αυτή. Διαφορετικά διατρέχουμε τον κίνδυνο να καταστρέψουμε κάποια από τα βασικά στοιχεία τη ευρωπαϊκή κοινωνία. Και κάτι άλλο. Νομίζω ότι στα έγγραφα των εμπειρογνωμών είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε περισσότερους εργαζόμενου. Η δημογραφική κρίση μα υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να δώσουμε Ευκαιρίε στι γυναίκε, όχι λόγω δικαιωμάτων, αλλά επειδή τι χρειαζόμαστε ή στου άνω των 50 ετών εργαζόμενου, όχι επειδή έχουν δικαίωμα μόνο, αλλά επειδή θα του χρειαστούμε στην αγορά εργασία. Στου μετανάστε, όχι επειδή είναι ανθρώπινα όντα, αλλά επειδή του χρειαζόμαστε για το κράτο πρόνοιας. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, όταν μιλάμε για τις γυναίκες, όταν μιλάμε για τους ηλικιωμένου εργαζόμενους, όταν μιλάμε για τους μετανάστες, να θυμόμαστε ότι όλους αυτούς τους χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε το συνταξιωτικό σύστημα. Όταν μιλάμε για την ε, ημέρα, για την, ε, συγγνώμη, για την αγορά εργασία, όταν πώς θα επιτρέψουν στις γυναίκες και στους υπόλοιπους να ενσωματωθούν σε αυτή την αγορά εργασίας όταν μιλάμε για εργασία χωρίς όρια. Πώ θα επιτρέψουμε την σωμάτωσή του στην αγορά εργασία, αν δεν του επιτρέψουμε να ασχοληθούμε με τι οικογένειέ του. Πώ θα επιτρέψουμε στου μετανάστε να ενταχθούν στην αγορά εργασία, αν δεν έχουμε τι απαραίτητε οδηγίε και δεν του δώσουμε κοινωνική πρόνοια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εδώ κάποια λογική, κάποια συνέπεια. Γι' αυτό ακριβώ, ε, Πρόεδρε, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα περίπλοκο εργαλείο. Με ένα εργαλείο αρκετά προχωρημένο, επειδή η κοινωνία μας είναι προχωρημένη. Κάποιοι λοιπόν έρχονται με κάποιες συνταγές πολύ απλές. Ζητώ από τους ε, συναδέλφους, γι' αυτό σημαντικό φάκελο, επειδή εγώ πιστεύω πολύ στην εργασία της εισηγήτριάς μας, ο φάκελος αυτός, η εισηγήση αυτή, αποτελεί μια ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι θέμα μόνο λογιστικής και θέμα πόρων. Το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Ευχαριστώ. Um, Mrs. Moran, followed by Mrs. Cornelison. Μωράν και μετά Κορνέλισεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την συγκήτρια Όμεν Ρόιτεν που επεξεργάζεται τα θέματα αυτά πολλά χρόνια εδώ στο Κοινοβούλιο, τα γνωρίζει καλά και κατάφερε να μας δώσει και τις γνώσεις της και την απαραίτητη στάθμιση που πρέπει να υπάρξει μεταξύ των διαφόρων απόψεων. Επίσης ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που μας ανέφεραν τις αναλύσεις τους και μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια πρόοδος στο θέμα των συντάξεων ακούγοντας διάφορες απόψεις και αναλύσεις μεταξύ συνδικάτων, Business Europe, όλα όσα ακούσαμε. Γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις διάφορες απόψεις για να προχωρήσουμε. Συμφωνώ με τον Αλεχάνδρο Σέρκας ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να είναι αντικείμενο πολιτικής διαμάχης πρόσκαιρης. Βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία και σήμερα ενώ συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση και μάλιστα βιώσιμη έτσι ώστε το σύστημα να μπορέσει να διαρκέσει πολλά χρόνια είναι τρομακτικό να θεωρούμε ότι μπορεί ένα τέτοιο θέμα τόσο σοβαρό, τόσο σημαντικό για την φιλοσοφική και οικονομική μας θεώρηση της κοινωνίας να το αντιμετωπίζουμε ως ε, θέμα πολιτικάντικο. Όπως είπα, η σύγκριση των διαφόρων συστημάτων είναι κάτι που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τα 27 κράτη-μέλη, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και εδώ πάλι η έκθεση της Ρίας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έλεγα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια οικονομία, μια φιλοσοφία αλλά και τις βαθιές αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Θα αρχίσω από τη φιλοσοφία μας η οποία είναι η αλληλεγγύη με το συνταξιοδοτικό σύστημα, το συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται σε μια αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών με ό,τι σημαίνει αυτό γενικότερα επί της οικονομίας. Και για την οικονομία θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να αρκεστούμε στη διαπίστωση του ότι όλο και αργότερα μπαίνουν οι νέοι στον κόσμο της εργασίας και από την άλλη να ζητάμε να μειώνεται ο χρόνος της εργασίας γιατί έχει ήδη μειωθεί πολύ και έτσι μειώνεται η συμβολή των εργαζομένων στον πλούτο μιας χώρας. Ξέρω ότι ο Θωμάς Μαν ασχολείται με το θέμα αυτό, την εργασία των μεγαλύτερων. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το θέμα της εργασίας των πιο ηλικιωμένων με τις, από τις συντάξεις. Πρέπει όμως να δούμε επίσης το ότι βρισκόμαστε στα μέσα κρίσης και ότι οι αποφάσεις των χωρών μελών πρέπει να λάβουν υπόψη τους και το θέμα των προϋπολογιστικών τους προβλημάτων. Τα οικονομικά προβλήματα της κάθε χώρας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε το πρόβλημα των συντάξεων. Σήμερα πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε στα ουσιώδη, δηλαδή να κρατήσουμε την ιδέα της αλληλεγγύης, αλλά με διαφοροποιήσεις. και μεταξύ των γενεών και του τρόπου που εργάζονται και μεταξύ των διαφόρων συνταξιδοτικών συστημάτων. Πολύ καλά το συνόψισε η Ρία στα πέντε της σημεία. Διασφάλιση επαρκούς σύνταξης που θα καθορίζουν τα κράτη-μέλη, διευκόλυνση της εργασίας και της σύνδεσης μεταξύ εργασίας και σύνταξης, κατάργηση των φραγμών προς την εργασία στις διάφορες χώρες μέλη, γιατί η ανεργία είναι πραγματικό πρόβλημα που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα και τέλος διάσωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων με περισσότερη διαφάνεια παρά την κρίση έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να έχει λογικά και αξιοπρεπή εισοδήματα για τη σύνταξή του. Η οικονομική κρίση μας οθεί να επιδείξουμε περισσότερη φαντασία και να συνδυάσουμε διάφορους και διαφορετικούς τρόπους εισφοράς και συνταξιοδότησης. Όχι ένα μόνο και ενιαίο σύστημα, αλλά πολλά συνδυασμένα. Η κινητικότητα των εργαζομένων που ενθαρρύνουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας υποχρεώνει επίσης προς τα εκεί να κινηθούμε. Σας ευχαριστώ. η κυρία Κορνέλισεν και μετά ο κύριος Μάν. Ευπρός η ευκαιρία ανταλλαγής με τους κοινωνικού εταίρους απόψεων για αυτό το σημαντικό φάκελο και έχω τρεις ερωτήσεις. Μετά από τα σχόλιά σας διερωτώ με πόσο μακριά πήγαν οι εργοδότες και τα συνδικάτα στις επαφές τους για να, για να συμφωνήσουν τελικά γιατί νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και αντιρρήσεις μεταξύ τους. Δεύτερη παρατήρηση σε σχέση με την ηλικία συνταξιδότησης. Είπαν όλοι την γνώμη τους. Νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να γίνει αυτό το θάμεο. Αυτό που με παραξενεύει όμως είναι το ότι πάντοτε αφορά μία αύξηση του ορίου ηλικία. Κανείς δεν φαίνεται να συζητάει ή να προβλέπει τη δυνατότητα προσδιορισμού του αριθμού ετών που, χρειάζεται, που χρειάζεται να δουλέψουν οι εργαζόμενοι. Γιατί αυτό θα ήταν πολύ πιο δίκαιο για τα άτομα που κάνουν σκληρότερες εργασίες και έχουν λιγότερα προσόντα και που ξεκινάνε νωρίς την εργασία τους και είναι σε ηλικία πανεπιστημικής μόρφωσης, ξεκινά δηλαδή 10-15 χρόνια πριν. Διερωτώ μου λοιπόν γιατί δεν το την υπόψη σας αυτό. Μετά. Όπως και αν το διοργανώσουμε αυτό, θα πρέπει να συνοδεύεται από την καταπολέμηση διακρίσεων λόγω ηλικία και με παραξενεύει το γεγονό ότι κανεί δεν το ανέφερε. Πολλοί άνω των 45 δεν μπορούν να βρουν δουλειά επειδή οι εργοδότε θεωρούν ότι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι μη παραγωγικοί και ότι ασθενούν συχνά. Στην Επιτροπή αυτή αναφέραμε μια Ολλανδική μελέτη που δείχνει το 80% των εργοδοτών δεν θα ήθελαν να προσλάβουν κανένα άνω των 40. Ήδη τα 40, από τα 40 και μετά θεωρήσε γέρος όσον αφορά την εργασία. Θα έπρεπε λοιπόν η Ένωση να καταβάλει προσπάθειες για την καταπολέμηση της αύξησης του ωραίου και θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να βρει ένα τρόπο μόχλευσης και για πίεση προς τις χώρες μέλη και τους εργοδότες για την διατήρηση και διασφάλιση των θέσεων εργασία, αλλά και για την επένδυση στην καταπολέμηση της διάκρισης λόγω ηλικία. Νομίζω ότι δεν γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την αλλαγή της στάσης των μελών των συνδικαλιστικών, των εργοδοτικών οργανώσεων για την αλλαγή της νοοτροπίας αυτής. Διαφορετικά δεν θα έχουμε και πάρα πολλούς στον χώρο εργασίας και θα έχουμε μεγάλη αύξηση του αριθμού των ανέργων και όχι του αριθμού των ατόμων που εργάζονται. Και ό,τι εξοικονομούν από τις συντάξεις οι χώρες μέλη θα τα δαπανίσουν μετά στα επιδόματα ανεργίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριος Μάν. Ευχαριστώ όλες. Είχα προετοιμάσει μια έκθεση για την Επιτροπή Απασχόλησης όσον αφορά την ε, δίκαιη κατανομή μεταξύ των γενιών που είχε μεγάλη επιτυχία γιατί έλαβε υπόψη τις προτάσεις όλων των συναδέλφων. έχουμε με αυτή μια καλή βάση. Αυτό χρειαζόμαστε. Σεβασμό μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων. Ο η συνάδελφος να αναφέρθηκε στις διακρίσεις. Αυτό δεν επιτρέπεται πια να υπάρχει και υπάρχει φαίνεται κάποια κίνηση. Η εφημερίδα Frankfurt Allgemeine της ε, Κυριακής είχε γράψει στον τίτλο της ε, την περισμένη εβδομάδα φαίνεται τελειώνει αυτή η λατρεία του νέου. Δηλαδή δεν θα λέμε ότι αρκεί να είναι κανένα νέος για να μπορέσει να είναι ο καλύτερος των αντίων. Οι πιο μεγάλη ηλικία έχουν πάρα πολλέ γνώσει, πάρα πολλέ ικανότητε και μπορούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πολύ καλύτερα. Και είχαμε πει ότι εντάξει, σα θέλουμε. είχαμε τους διάφορους δικούς σας εκπροσώπους που είπαμε τι γίνεται με αυτές τις θέσεις απασχόλησης στις οποίες συνεργάζονται οι νέοι και οι ηλικιωμένοι συγκεκριμένα. Δηλαδή από κοινού, κοινό έργο και ε, συνένωση των εμπειριών των άλλων. Ευτυχώ υπάρχουν όσο πάει και πιο συγκεκριμένε προτάσει για το τι θέλουμε να αλλάξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα. Δεύτερον, τι θέλουμε. Θέλουμε οι νέοι να μπουν στην αγορά απασχόλησης γιατί έχουν πραγματικά τα απαραίτητα προσόντα. Έχουν τις προϋποθέσεις για να μπορούν να εργαστούν και να εργαστούν και για πιο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό θέλουμε. Δεν μπορούμε να τους πούμε ότι θα πρέπει πιο γλίγορα να μπείτε στην αγορά απασχόλησης γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει το θέμα των προσόντων. Θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται κανένας μία μακροχρόνια εκπαίδευση για να μπορέσει να ε, αντιμετωπίσει τις ανάγκες της αγοράς. Δεν μπορούμε να το αποχωρήσουμε αυτό. Θέμα αρχή τώρα. Αυτή η πράσινη βίβλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, υποβάλλουμε μόνο ερωτήσεις. Αλλά με μια σειρά ερωτήσεων δίνει τη δυνατότητα ότι κάτι, η ιδέα συγγνώμη, ότι κάτι άλλο πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, δεν ε, πρέπει να έχουμε εδώ πέρα μία αίτηση σαν ε, να υπάρχει δηλαδή κοινοτική αρμοδιότητα. Όλοι θα πρέπει να παραμείνουν, όλα τα θέματα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εάν αυτό είναι σημαντικό για ένα κοινό μήνυμα, εντάξει. Να πούμε δηλαδή, έχουμε στα κράτη-μέλη ανεξάρτητα συστήματα συνταξιοδότηση και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα σχετικά κριτήρια. Δεν θέλουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα ηλικία συνταξιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αναφέρθηκε ήδη τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Γαλλία. Ε, τελικά θα περάσουν από τα 65 στα 67, όπως το έχουμε και στη Γερμανία. Και τέλος, χρειαζόμαστε μια ενιαία περιγραφή του επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος κράτη-μέλη ρωτάνε γιατί ασχολείται η Ευρώπη τόσο πολύ. Ε, όταν βλέπω ότι έχουμε μεταξύ 2 και 4% των πολιτών που λένε ότι έχουμε μια απασχόληση σε ένα κράτος μέλος στην αρχή και μετά σε μια άλλη χώρα μέλος. Λοιπόν, τα αριθμητικά στοιχεία είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Δεν οφείλεται στο γεγονό ότι έχουμε διαφορετικά συνταξιδοτικά συστήματα, αλλά ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητα. Και ένα σημείο που για μένα είναι επίση σημαντικό είναι οι ε, ιδιωτικέ ε, επαγγελματικέ συντάξει από τι επιχειρήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και αυτό σχετίζεται με αυτό που είπαμε για το θέμα της μεταφοράς τα τελευταία χρόνια. Ορισμένοι συνάδελφοι από τη δική μας Επιτροπή και άλλες, πολλοί δεν ήξεραν γιατί στη Γερμανία έχουμε τόσο μεγάλη εμπειρία και επιτυχία με αυτά τα συστήματα των ε, επιχειρησιακών συντάξεων. Γιατί στη Γερμανία επιβραβεύονται οι εργαζόμενοι όταν παραμείνουμε στην ίδια εταιρεία. Δεν είναι θέμα ε, κινητικότητας που λέμε, όχι. Είναι σημαντικό κριτήριο το να έχει παραμείνει κανένας στην ίδια επιχείρηση. Και αυτό δεν είναι κάτι που βοηθάει να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Λοιπόν, ευρωπαϊκές συμβολές ναι, καλό. Θέλουμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Καλό. Θέλουμε η εμπειρία των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων να ληφθεί περισσότερο υπόψη στα κράτη-μέλη. Και τέλος, είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, επικοινωνούμε για τις διαφορές αυτές. Αλλά βέβαια με ξεκάθαρα λόγια όχι σαν τους, ε, αυτούς που απλώς συζητάνε για παραγράφους. Όχι, μια ευγνώτη γλώσσα γιατί νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Αν δηλαδή, Λίζ, έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, θέλουμε να φροντίσουμε η αρμοδιότητα να μείνει στα κράτη-μέλη, από εκεί και πέρα όμω μπορούμε να κινηθούμε. Αυτά είναι καλά. Και όχι να πούμε ότι θα έχουμε ε, μια ευρωπαϊκή κάλυψη πάνω από όλα. Αυτό δεν θα ήταν σωστό μήνυμα. Uh, ευχαριστώ, Χάκιν και μετά κύριε Φιγκερέντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο Τόμας Μαν το ξεχθάσε το θέμα και να ευχαριστήσω την συγγύτρια καταρχήν για τη θαυμάσια δουλειά τη. Πολύ καλή ιδέα να έχουμε τους κοινωνικούς εδώ σήμερα και ευχαριστώ για τις συμβολές τους επειδή ακριβώ διευρύνει τον ορίζοντα των σκέψεων και των επιχειρημάτων και εμπλουτίζει την εμπειρία μας. Σε αυτά που έλεγε ο Τόμας Μαν και που ανέφεραν και άλλοι ομιλητές σήμερα εδώ, το θέμα της επιρικότητας και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι δύο πράγματα που αντιμετωπίζουμε κυρίως μέθοδο συντονισμού και πολλοί είπαν και συμφωνώ ότι θα πρέπει να δούμε τα θέματα της καταλληλότητας, ηλικίας κτλ. Και αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί σε επίπεδο χώρας, μέλους. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε εδώ και άλλα επιχειρήματα. Νομίζω ότι περισσότεροι συμφωνούμε για αυτά τα θέματα. Όμως έχουμε και το δεύτερο ζήτημα, η σταθερότητα. Η σταθερότητα του ευρώ τα δημόσια οικονομικά και διασφάλιση των συντάξεων. Χθες, στην αρχή της ε, συνεδρίασης, δεν ήμουν εδώ και μιλήσατε για αυτά τα θέματα νομίζω. Να κάνω και ένα σχόλιο εδώ, ότι εδώ κατάγω μια χώρα, την Ιρλανδία, που αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες και θα είναι αδύνατο να ακολουθήσουμε τις επιταγές του Συμφώνου Σταθερότητας μέχρι το 2014. Το σύμφωνο βεβαίω είναι σημαντικό για τα δημοσιοοικονομικά, αλλά δεν θα ήθελα η συζήτηση αυτή να μπλεχτεί με τι ημερομηνίε για το μέχρι πότε θα πρέπει οι χώρε μέλη να εφαρμόσουν τι επιταγέ του Συμφώνου Σταθερότητα. Για του κοινωνικού εταίρου και τα θέματα που συζητήθηκαν, έχω κάποιε ερωτήσει που θα ήθελα να σα θέσω. Καταρχήν, Business Europe. εσεί μιλήσατε ότι δεν χρειάζεται αναθεώρηση της οδηγίας και επιχειρηματολογήσατε λέγοντας ότι η Κομισιόν βρίσκεται υπό διαβούλευση και αναζητά απαντήσεις. Να ρωτήσω, αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο θεωρείτε ότι δεν χρειαζόμαστε αναθεώρηση της οδηγίας, επειδή βρισκόμαστε μόνο στην διαδικασία αναθεώρησης δεν χρειάζεται, νομίζετε, καθόλου αναθεώρηση. Δεύτερον, διαφοροποίηση πόρων όσον αφορά τα κονδύλια για τι ε, συντάξει κάτι που έθεσαν και άλλοι ομιλητέ. Ποιε ιδέε έχετε για αυτό το θέμα, ποιου άλλου πόρου προβλέπετε οι πηγέ κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των συνταξιωτικών ταμείων. Αναφερθήκατε όπως και άλλοι ομιλητές για συμπληρωματικούς κανόνες φερεγγιότητας. Για τους περισσότερους ομιλητές φαίνεται ότι αυτό δεν χρειάζεται. Να ρωτήσω, θα πρέπει να υπάρχει μια πιο συστηματική νομοθεσία για τις συντάξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι γίνεται με τις δικλείες ασφαλείας που θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε για να μειώσουμε τους κινδύνους. Και αυτό το ερώτημα αφορά όλους τους κοινωνικούς εταίρους, γιατί το ανέφεραν επανειλημμένως κι άλλοι. Η ETAC, τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, Κάποια από τα αρχικά σα σχόλια ήταν το ότι δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούμε τη γύρανση του πληθυσμού. Δεν νομίζω θα συμφωνήσω γι' αυτό που λέτε. Αν δείτε τα στοιχεία ο αριθμός των ατόμων που σταξιοτέθηκε από το 97 και μετά διπλασιάστηκε και από το 2012 θα μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ λοιπόν να συμφωνήσω μαζί σας ότι υπερεκτιμάμε το θέμα του αντίκτυπου της γύρανσης και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε αυτό. Μιλήσατε επίσης για το ότι η προτεραιότητά σας είναι η ποιότητα της εργασίας και η ποιότητα των αμοιβών. Νομίζω ότι αυτό σε γενικέ γραμμές είναι και η δική μας προτεραιότητα. Να ρωτήσω όμως το εξή. Πόσο συγκεκριμένα θα συνδέατε εσείς την ποιότητα των αμοιβών και την ποιότητα των, της εργασίας με το θέμα των κατάλληλων και των βιώσιμων συντάξεων. Θα ήθελα να αποψή σας από αυτού. Να ρωτήσω και το εξής και δεν νομίζω να το άκουσα εδώ, για το αναδιονομητικό στοιχείο της σύνταξης. Δηλαδή σύνταξη που συνδέεται με, τις, με τα εισοδήματα και σύνταξη η οποία βοηθάει τους ηλικιωμένου να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Αναφέρθηκε ένα σχόλιο για την πρόορη ταξιδότηση. Και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι πριν από λίγους μήνες είδαμε ποιες χώρες μέλη ανταποκρινόταν στην οικονομική κρίση και κάποιες οικονομικές χώρες, κάποιες χώρες συγγνώμη, μέλη, όπως η Σουηδία, Δανία ενδεχομένω, Γερμανία, έκανα μια σύνδεση της πρόορης δαξιδότησης και της πρόσληψης νέων ατόμων και ένταξή του στην αγορά εργασία. Κατανοώ αυτά που λέτε για την πρόορη δεξιοδότηση. Όμω, μήπω αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ω μηχανισμό για την πρόσληψη περισσότερων νέων ατόμων. Θέλω σχόλια από αυτού. Επίσης έγινε λόγος για ένα πλαίσιο και μια ανάμειξη λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις λύσεις που ακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα τι εννοείτε με αυτό. Κατανοώ αυτό που λέτε, αλλά δεν έχω αντίληψη των λεπτομεριών που αναφέρατε εσείς. Και τέλος, κάποια γρήγορα σχόλια να κάνω. Να σας πω το εξή: Όλοι μιλάνε για παράταση της σταδιοδρομίας και του χρόνου της εργατικής ζωής των εργαζομένων. Όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο της μείωσης του χρόνου εργασίας, το ρόλο της τεχνολογίας εδώ και το θέμα των πόρων που θα χρειαστούν για την χρηματοδότηση των συνταξιδοτικών ταμείων. Θα ήθελα να μιλήσω επίσης και για το θέμα της πρόνοιας, της άτυπης πρόνοιας. Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Αυτοί που παρέχουν ένα είδος άτυπης πρόνοιας, ιδιαίτερα σε πλαίσιο οικογενειακό, πολύ συχνά όταν φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης έχουν χαμηλότερες συντάξεις. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτά τα άτομα. Επίσης, για την ανάγκη υποστήριξης της άτυπης πρόνοιας. Επειδή ο κόσμος ζει περισσότερο, οπότε η άτυπη πρόνοια είναι σημαντική και επιμικύνεται χρονικά. Δύο επίσης θέματα σημαντικά. Το θέμα του φίλου Επειδή οι γυναίκες σταξιδοτούνται νωρίτερα από τους άντρες. Για το 2007 είχαμε διαφορά γύρω στα δύο χρόνια. Και όταν έχουμε ε, συνταξιοδότηση με χαμηλότερε συντάξει, θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό είναι θετικό ή όχι. Και μια ερώτηση προ όλου του εταίρου. Μήπω θα έπρεπε η κάθε γενιά να βασίζεται στην νεότερη γενιά για τη χρηματοδότηση των συντάξεων ή μήπω εναλλακτικά θα έπρεπε να κοιτάξουμε άλλου τρόπου χρηματοδότηση των συντάξεων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έδωσε ένα συγκεκριμένο ορισμό των συντάξεων. Συντάξεις με αυτό τον ορισμό του δικαστηρίου ή συντάξεις όπου η νεότερη γενιά χρηματοδοτεί την προηγούμενη γενιά. Έχετε κάποια άποψη για αυτές τις δύο ε, περιπτώσεις ή προβλέπετε να συνδέσουμε και το δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Άρκιν έθεσε πάρα πολλά ερωτήματα και νομίζω ότι κάλυψε πάρα πολλές πτυχές του θέματος μας. Εγώ θα ήθελα αντίθετα να επικεντρωθώ σε τρία σημεία. Ένα πρώτο ζήτημα ουσίας είναι το εξής. Είναι το να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που θα επιτρέπει σε όλα τα άτομα σε όλους τους ανθρώπους να ζουν μια ζωή αξιοπρεπή. Ιδιαίτερα σε περιόδους της ζωής τους όπου δεν θα εργάζονται. Και αυτό το δημόσιο σύστημα θα πρέπει, δημόσιο σύστημα πρόνοιας, θα πρέπει να συνοδεύεται από άλλες μορφές ή πηγές χρηματοδότησης. Γιατί βλέπουμε ότι το δημόσιο σύστημα πρόνοιας χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται βασιζόμενο στις εισφορές των εργαζομένων και χρησιμοποιείται όχι μόνο για να γίνονται και να διασφαλίζονται οι μεταρρυθμίσεις, αλλά και για να διασφαλίζεται μια πολιτική απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους. Το θέμα των προκατακτικών μεταρρυθμίσεων. Ενδεχομένως ε, χρησιμοποιείται και για την χρηματοδότηση της ε, κατάρτισης. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτούνται και τα επιδόματα ανεργίας. Σε τελική ανάλυση λοιπόν, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής πρόνοιας αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Οπότε μας λένε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το όριο θα πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο. Διαφορετικά, τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα ύπαρξης στο μέλλον. Το θέμα λοιπόν ουσία είναι το εξή. Γιατί θα πρέπει να διακρίνουμε το σύστημα μεταρρύθμιση βάσει των εισφορών των εργαζομένων, να το διακρίνουμε δηλαδή αυτό από την στήριξη της κοινωνικής πρόνοιας η οποία θα πρέπει να ισχύει για όλους βάσει ενός συστήματος που δεν θα βασίζεται στις εισφορές. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρες μέλη μέσω του προϋπολογισμού τους να καλύπτουν αυτές τις ε, περιπτώσεις και μιλάω ας πούμε για την ύπαρξη ενός ελάχιστου εισοδήματος που θα πρέπει να υπάρχει και να είναι διαθέσιμο σε όλους ώστε να καταπολεμήσουμε την φτώχεια και να επιτρέψουμε στα παιδιά μας και στους νέους μας να ξεφύγουν από την φτώχεια η οποία αφισβητεί το μέλλον τους για να μην ε, θέσουμε σε ένα αμφιβόλο μάλλον το μέλλον των ε, επερχόμενων γενεών. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συγχέουμε τα συστήματα εισφορών με τα συστήματα που δεν περιλαμβάνουν εισφορές. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα το οποίο βασίζεται σε εισφορές θα πρέπει βεβαίως να καταβάλει επιδόματα από τα συστήματα τα οποία δεν προβλέπονται από τα συστήματα που δεν βασίζονται στις φορές όπως το, όπως το ε, χαμηλότερο εισόδημα. Δεύτερο ζήτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Η επιμέκυνση της ζωής των εργαζομένων δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα είδος τιμωρίας για τους εργαζόμενους τους ίδιους. θα πρέπει να βρούμε τρόπους αντίθετα βελτίωσης των συνθήκων ζωής. Τη στιγμή που μάλιστα που σήμερα έχουμε επιμήκυνση της ζωής ή του ορίου ζωής και το προσδόκιμο ζωής ε, φτάνει πια τα 80-82 έτη. Όμως αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν έγκλημα λόγω του οποίου θα πρέπει να τιμωρήσουμε δηλαδή τους εργαζόμενους επιμικίνοντας τον χρόνο εργασίας. Συμφωνώ με την κυρία Άρκιν λοιπόν και τα σχόλιά της για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα. Η τεχνολογία θα πρέπει να μας επιτρέπει να κάνουμε βελτιώσεις. Βελτιώσεις για όλους, δηλαδή να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, να έχουμε μικρότερο χρόνο εργασία, περισσότερο χρόνο για την κατάρτιση, περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μας κλπ. κλπ. Οπότε, πού βρίσκεται αυτό το θετικό στοιχείο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και το τρίτο ερώτημα που έχω να θέσω αφορά το μέλλον των νέων. Επειδή αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση παρατείνεται η, η παρουσία των εργαζομένων στην αγορά εργασίας αυτό θα έχει ως συνέπεια την μικρότερη ή τη χαμηλότερη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και αυτό θα θέσει κίνδυνο το, το μέλλον τους. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι οι αγώνες και όλες οι διαμαρτυρίες που έχουμε στις διάφορες χώρες μέλη κατά της αύξησης του ορίου ηλικίας αποτελούν στην ουσία μία προάσπιση και μία υποστήριξη των μελλοντικών γενεών και κυρίως των νέων. Και αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα νομίζω εδώ. Και πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε μια καθαρά φιλελεύθερη και οικονομικιστική προσέγγιση, κατά κάποιο τρόπο υποθηκεύουμε το μέλλον. Ε, και κατά συνέπεια κάνουμε υποχωρήσεις όσον αφορά τις κατακτήσεις και τα επιτεύγματα του πολιτισμού, γιατί θα οδηγηθούμε σε προβλήματα φτώχεια, σε διακρίσει σε μείωση του προσδοκιμού ζωή και μείωση τη ποιότητα τη ζωή. και αυτό ήδη το έχουμε δει. Επαντλημένος λοιπόν θεωρώ ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθήσει αυτό το δρόμο θα καταλήξει ακριβώς αυτή την κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε είναι μεγάλη σημασία και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα ήθελα να σα παρουσιάσω αυτέ τι ανησυχίε μου και τι απόψει μου όσον αφορά τις ε, απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα τεκτονόμενα στις διάφορες χώρες μέλη. Νομίζω ότι το θέμα είναι ξεκάθαρα θέμα επικουρικότητας, αλλά νομίζω είναι εξίσου ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις μακροοικονομικές πολιτικές που επιβάλλει στις χώρες μέλη όπως η αυστηρή τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ακριβώς συμβάλλει σε μια ενίσχυση των διακρίσεων και των διαφορών και σε μια αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, εάν και εφόσον υπήρξε ποτέ αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Φιγκερίντο. Άσχημα νέα, οι επόμενοι ομιλητέ θα έχουν λιγότερο χρόνο. Γιατί μου λένε ότι καθυστερήσατε πολύ. Ή μάλλον να πω ότι χρησιμοποιήσατε πολύ χρόνο. Λοιπόν, κύριε Άγγελ, λυπούμε που θα είστε ο πρώτος με το λιγότερο χρόνο, αλλά παρακαλώ κάτω των δύο λεπτών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καθώς και για τις περιορισμούς που επιβάλλατε. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη άλλοι τα προβλήματα. Πρώτον, η εργασία φαίνεται ότι ενοχλεί πολλούς γιατί δεν τους αφήνει αρκετό ελεύθερο χρόνο. Δεύτερον, φαίνεται ότι από το πέρασμα της φοιτητική ζωής στη σύνταξη πολλοί θέλουν το ενδιάμεσο διάστημα να μειωθεί ως το δυνατόν περισσότερο. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω πώς άρχισε το συνταξιοδοτικό σύστημα. Ήταν ασφαλιστικό κατά του κινδύνου τότε λίγο πιθανού να φτάσει κανείς σε ηλικία όπου να μην μπορεί πια να δουλέψει. Τώρα όμως έχουν, έχει γίνει η σύνταξη ο άλλος τρόπος ζωής επί πολλές δεκαετίες. Και υπάρχει λοιπόν εδώ το δημογραφικό πρόβλημα. Ξέρω ότι δεν συμφωνούν οι περισσότεροι μαζί μου, αλλά τίθεται και το βασικό πρόβλημα εδώ ότι χρειάζεται όλο και περισσότερος χρόνος για την κατάρτιση και πολύ συχνά 25 και 30 χρόνια εργασίας δεν αρκούν για να χρηματοδοτήσουν ακόμη τόσα χρόνια σύνταξης. Στο Λουξεμβούργο υπολογίζεται ότι 16% του ΑΕΠ αφιερώνεται στη χρηματοδότηση των συντάξεων. Και αυτό θα έπρεπε να ανησυχήσει και τις επόμενες γενιές. Όλο θέμα επικουρικότητας και ξέρω ότι πρέπει να παραμείνουν όλα αυτά εθνικό θέμα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων αν δεν υπάρξει και μεγαλύτερη συγκρισιμότητα και συνδυασμός των συστημάτων συνταξιοδότησης. Αυτό μου φαίνεται τελείως βασικό. Χιλιάδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα γιατί έχουν εργαστεί σε δύο-τρία διαφορετικά μέρη, διαφορετικές χώρες και ο συνδυασμός των δικαιωμάτων είναι πολύ δύσκολος ακόμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Νταρντέν και μετά ο κύριος Κονφεράτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώνουμε σήμερα πόσο πλούσια είναι αυτή η συζήτηση και πόσο διαφορετικές οι απόψεις. Το θέμα είναι πολύπλοκο και είναι σημαντικό να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Γιατί πρόκειται για πραγματικά κοινωνικό θέμα και θα επανέλθω σε μερικά, μερικές από τις πτυχές του για να εκφραστώ προσωπικά. Πρώτον, ο ρόλος της Ευρώπης. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε στη λογική της επικουρικότητας. Αλλά δεν θα έπρεπε να περιοριστούμε σε αυτό. Γιατί το θέμα αυτό που κινητοποιεί τον κόσμο παντού στην Ευρώπη και που είναι και επίκαιρο αλλά και αφορά και το μέλλον πρέπει να έχει κάποια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Χωρίς αυτήν πώς μπορεί να υπάρξει μία συνεπής πανευρωπαϊκή στάση. Πρέπει λοιπόν κάποια συνοχή. Πρέπει να ξεπεράσουμε το απλό θέμα του ποιες ακριβώς είναι οι δικαιοδοσίες της Ένωσης και να μπούμε σε μια λογική συντονισμού, ενισχυμένου συντονισμού των προγραμμάτων μας. Δεύτερον, η σημασία των πυλώνων. Είναι σαφές ότι όλοι οι πυλώνες είναι χρήσιμοι και συμπληρωματικοί ο ένας με τον άλλον, αλλά επίσης βασικό είναι να κρατήσουμε έναν ισχυρό δημόσιο πυλώνα γιατί αυτός θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη εγγύηση της αλληλεγγύης και κάποια ασφάλεια των συντάξεων. Επ' αυτού πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα στην αλληλεγγύη γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια σταδιοδρομία, τις ίδιες διευκολύνσεις, την ίδια πρόσβαση στην εργασία και άρα ιδιαίτερα οι άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες και πρέπει να παραμείνει σημαντικός αυτός ο πυλών. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ηλικία της συνταξιοδότησης. Γίνεται πολλής λόγος, ακούγονται διαμάχες. Μερικοί λένε ότι η αγορά της εργασίας δεν καταλήγει σε απλή εκαθάριση και εκμηδενισμό, πρέπει να παραλληλήσουμε την ηλικία της συνταξιοδότης, την ποιότητα της εργασίας και να συνδυάσουμε καλύτερα την πραγματική ηλικία συνταξιοδότης με την νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης. Τέλος, κοιτάξτε, αν μιλήσετε όλοι όπως ο κύριος Αγγέλ, ε, καταλαβαίνω ότι το θέλετε, αλλά δεν θα προλάβουν όλοι. Τέλος, το ποσό της σύνταξης. Κατανοώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει ενιαίο ποσοστό ευρωπαϊκό, αλλά κάποιο ελάχιστο ποσοστό θα μπορούσε να καθοριστεί πανενοσιακά, όπως είχαμε μιλήσει για το ελάχιστο εισόδημα, για να μπορέσουν οι ηλικιωμένοι να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή στη σύνταξή τους. Ο κύριος Κοφεράτη και μετά ο κύριος Βαλτασάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι στο θέμα των συντάξεων ο ρόλος Ευρώπης είναι πολύ σημαντικός. Δεν με την άποψη ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να αφηθούν, να αφαιθούν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα πρέπει να υπάρχει νομίζω ένας προσανατολισμός και θα πρέπει να υπάρχει μια νέα δομή για την Ευρώπη. Όταν για ένα άτομο μιλάμε για κράτος ευημερίας, τότε η πλειοψηφία των πολιτών έχει κατά νου τις συντάξεις, ένα από τα κυριότερα στοιχεία του κράτους ευημερία. Βεβαίως και οι δημογραφικές εξελίξεις ε, μας υποχρεώνουν να λάβουμε υπόψη μας κάποια πράγματα και να τα αντιμετωπίσουμε και να τα λύσουμε. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει που να ξεχάσουμε ή να παραβλέψουμε τον ουσιώδη ρόλο του δημόσιου πυλώνα. Θεωρώ όμως ότι μελλοντικά με τις αυξήσεις του ορίου ηλικίας στην Ευρώπη και με τη διαδικασία ταυτόχρονα της αύξησης του γυρότερου πληθυσμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία, τότε είναι αναπόφευκτο η κρατική πρόνοια να μην αυξηθεί ή να προσαρμοστεί αντίστοιχα σύμφωνα με τον αρχικό της ρόλο. Οπότε έχουμε το τρίτο πυλώνα. Τρίτο πυλώνα όπου όμως θα, έχουμε, θα πρέπει να έχουμε φορολογικά κίνητρα. Και είναι σημαντικό εδώ να κάνει κάποιες προσπάθειες η Ευρώπη όσον αφορά τον, τον προορισμό των κονδυλίων και την αναθεώρηση. Η κινητικότητα. Θα πρέπει να πούμε ότι για δημογραφικούς λόγους θα έχουμε εκατομμύρια μεταναστών στην Ευρώπη Οπότε το θέμα της κινητικότητας και της διαχείρισης των δικαιωμάτων τους αποτελεί ένα θέμα ουσιώδες όσον αφορά τα πολιτιακά ζητήματα. Ένα άλλο θέμα σημαντικό είναι η ευελιξία. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να εισάγουμε στα διάφορα προγράμματα ως βασικό δικαίωμα το δικαίωμα διάκρισης από εργασία σε εργασία και από συνθήκες εργασία σε συνθήκες εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν θα πάνε ε, στη σύνταξη ή αν θα παραμείνουν στην εργασία τους. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι ίδιες όλες οι δουλειές. Κάποιες ε, ε, ε χρειάζονται ενδεχομένως περισσότερη πρόνοια σε σχέση με κάποιες άλλες. ο κ. Παλτασάρ και μετά κυρία Στρέτερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το εύρος που έδωσε σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι η ιστορία των ευρωπαϊκών οργάνων μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες περιόδους νηνεμίας και μετά μια ξαφνική επιτάχυνση των θεσμικών ζητημάτων. Η τελευταία κρίση της Παρασκευής ε, το βράδυ όπου είχαν ληφθεί αποφάσεις που δεν προέβλεπαν οι συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι και σε αυτό το τομέα βρισκόμαστε νομίζω σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούμε να μείνουμε απλοί θεατές όσον αφορά την επικουρικότητα για τις χώρες μέλη και αποτελεί μια, νομίζω μια λογική συνέπεια της κατάστασης που αφορά την ίδια την Ευρώπη που έστω και δεν έχει αρμοδιότητες νομοθετικές θα πρέπει να δώσει κάποιες κατευθυντές γραμμές, γραμμές κάποιων προσανατολισμών. Δεν θα πρέπει να προβλέψουμε ή δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε 27 χώρες να υπάρχουν δημοσιονομικές πολιτικές διαφορετικές. Αυτό ήδη εναρμονίζεται. Οπότε αντίστοιχα θα πρέπει να έχουμε και πολιτικές συνταξιοδοτικές ομοιογενείς. Δεν γίνεται στη Γερμανία κανεί να συνταξιδοτείται στα 68 και αλλού στα 50. Αυτό το έχουμε δει. Και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να έχουμε κινητικότητα και ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων αν στις χώρες μετακίνησης των εργαζομένων δεν υπάρχουν και απαραίτητες εγγυήσει για την ασφάλιση του μέλλοντός τους. Καταρχήν λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα ένταξης στα ευρωπαϊκά συντοξιδοτικά συστήματα, όλο προηγουμένω ο συνάδελφος από το Λουξεμβούργο, η Ιταλοί, τα τελευταία χρόνια αποτελούσαν ένα σημαντικό ποσοστό της εσωτερικής μετανάστευσης και υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι που δούλεψαν στην Γαλλία, στην Γερμανία, στην Ελβετία και σε άλλες χώρες. Οπότε ο ελάχιστο στόχος εδώ είναι η ένταξη αυτών των θέσεων στα συστήματα εισφορών με, μια, με ένα ελάχιστον παρονομαστή. Πρόεδρε, καταλήγω. θέλω να πω ότι δεν γίνεται να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές ξεκάθαρες επειδή ακριβώς δεν είμαστε ακόμα σε θέση να πάρουμε μια ενιαία θέση για, την, για το όριο ηλικία. Υπάρχει μόνο μια συνολική λογική που επιβάλλει τέλο πάντων κάποια κριτήρια συνολικά για το όριο ηλικία. Δεν γίνεται όμως να έχουμε αποκλήσεις πολύ σημαντικές όσον αφορά την ίση μεταχείριση. Κανείς δεν, δεν μπορεί κανείς να αποδεχτεί ότι σε μια χώρα συνταξιδοτεί κανεί με το 70-80% του τελευταίου μισθού, ενώ σε μια άλλη χώρα γίνεται αυτό με το 40%. Και τελειώνω, Πρόεδρε, θα πρέπει να υπάρχουν ίδιες ε, συνθήκες ε, αγοραστική δύναμη σε όλε τις χώρες. Οπότε η απασχόληση και τα θέματα της ε, συνταξιοδότησης, όλα αυτά θα πρέπει να είναι εξίσου παρόντα στι κατευθύνσεις γραμμένε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, καταλαβαίνουμε πέρα τον πρόκειται. Το να υπάρχει ένα ελάχιστο ευρωπαϊκό λόγω των κρατικών ε, διαφορών ε, απ' την άλλη μεριά, αν θα πρέπει να, υπάρχει εκεί μια διακίνηση ανάλογα με την ηλικία στην οποία συνταξιοδοτούνται, ανάλογα με την σύνθεση, τη δημογραφική της ε, ε, χώρας αυτής, δεν μου φαίνεται σωστό. Η κυρία Σουέτερ, παρουσιάστε ένα καινούργιο επιχειρήματα. Εγώ όμως θέλω να αναφερθώ στο σύνολο της συζήτησης. Καταρχήν, το ερώτημα, γιατί η Κομισιό υπέβαλε αυτή την πράσινη βίβλο γιατί υποθέτω ότι θέλει να ε, φροντίσει να μπορέσει να κινητοποιηθεί η δυνατότητα, η δυνατότητα της μεταφοράς των συντάξεων. Αυτό είναι σωστό. Αυτό που χρειάζεται είναι η μεταφορά των συντάξεων να σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή θα αφαιρέσουμε χρήματα από τους ε, αφαιρούμε μάλλον χρήματα από τους εργαζόμενους γιατί δεν προωθούνται δεν έχει λυθεί το θέμα. Είναι προφανές ότι κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Δεύτερον, και εκεί θα μπορούσε να δράσει και η Κομισιόν, και ανεξάρτητα από την πράσινη βίβλιο, είναι ότι η καλή εργασία οδηγεί σε καλές συντάξει. Όσον αφορά δηλαδή τους ε, όρους εργασίας θα πρέπει να είμαστε πιο ε, δραστήριοι. Πάρα πολύ σημαντικό. Τρίτο σημείο το θέμα των διακρίσεων. Και εδώ έχει η η Κομισιόν και χρειάζεται νομίζω οι μεγαλύτερε ηλικίε ε, εργαζόμενοι να μπορέσουν ε, να συνεχίσουν να εργάζονται. Και αυτό προφανώ είναι ένα θέμα στο οποίο η Κομισιόν μπορεί να φροντίσει να εφαρμοστεί η σχετική οδηγία. Τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω είναι η δυνατότητα του ανοιχτού συστήματο συντονισμού, κάτι που γίνει και στο Συμβούλιο, και θα ήταν καλό να έχουμε ε, τις βέλτιστες πρακτικές και οι βέλτιστες πρακτικές μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές και όσον αφορά δημοκρατική ε, μετατροπή, χωρίς να περιορίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και εδώ θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε λύσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν στο μέλλον. Το κεντρικό θέμα όμως όσον αφορά τις δράσεις της Κομισιόν είναι η σημερινή κατάσταση. Και αυτά είναι τα τρία θέματα που σας ε, παρουσίασα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ ε, σύντομα και τηλεγραφικά. Στη διάρκεια της συζήτησης α, ε, υπόθηκαν πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Σημειώνω ότι ήταν εξαιρετική για μένα και συμφωνώ απολύτως με την εισήγηση του κυρίου Σέρκας περιέγραψε την κατάσταση έτσι ακριβώς όπως υπάρχει σήμερα και ταυτοχρόνως συμφωνώ απολύτως με τα ερωτήματα της κυρίας Χάρκιν για τα οποία και περιμένω απαντήσεις. Βάζω δύο ακόμα σημεία. Νομίζω ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει ευθύνη για δικές του αποφάσεις, αλλά ταυτοχρόνως θα ήθελα και ένα γενικό προσανατολισμό. Ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια εξαιρετικά πολύπλοκη κατάσταση. Βρισκόμαστε στην εξέλιξη μιας νομοθετικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της οποίας αυξάνουμε τα όρια ηλικίας στις συντάξεις. Μειώνουμε τα ποσά των συντάξεων, ενώ ταυτοχρόνως αυξάνεται η ανεργία. Την ίδια στιγμή καλούμαστε από την Ευρώπη να επιτύχουμε στόχους που αφορούν τα ζητήματα της απασχόλησης και της φτώχειας. Αντιλαμβάνεστε ότι για να τα κάνει όλα αυτά μια κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ταχυδακτηλουργικές ικανότητες. Γι' αυτό και χτες το βράδυ σε μια συνέντευξη σε πανελλήνιο δίκτυο του Πρωθυπουργού με αφορμή τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ετέθη το δίλημα ή θα στηρίξετε ως ελληνικός λαός αυτή την προσπάθεια που κάνουμε με όλες τις δυσκολίες ή θα πάμε στις εκλογές. Αναφέρω αυτό το ελληνικό παράδειγμα για να αντιληφθούμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να συγκεράσουμε όλα τα ζητήματα. Έχουμε μπροστά μας μία, εξίσωση με πάρα πολλές μεταβλητές. Υπάρχουν δύο τρόποι για να λυθεί. Ο ένας τρόπος είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε εδώ με ε, συζήτηση, με ανταλλαγή απόψεων και κυρίως με το να βρούμε έξυπνες λύσεις. Ο άλλος τρόπος, και το λέω ε, σκοπτικά, το λέω κάνοντας μαύρο χιούμορ και ε, μεταφέροντας την, κάτι που είπε ένας φίλος με πολύ μεγάλη εμπειρία στα πολιτικά ζητήματα, ο άλλος αυτός τρόπος είναι να προωθήσουμε την ευθανασία στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Δεν euh, φαντάζομαι να συμφωνώ πολύ. Κυρία Όμεν Ρόιτεν, θέλετε σε αυτήν τη φάση να ξαναμιλήσετε για να θέσετε κανένα ερώτημα στους εμπειρογνώμονες πριν τους ξαναδώσω το λόγο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις και τα σχόλια αυτά. Κυρία Εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μου πούν το εξής. Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων πώς μπορεί κανείς να φανταστεί ότι το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του. Αν θέλουμε επαρκή σύνταξη, κάτι που το δέχομαι, τότε τότε λέγω εδώ κάτι δεν κολλάει. Το καθαρό εισόδημα θα χαμηλώσει ή θα χαμηλώσουν οι εισφορές. Αυτό βέβαια θα έχει επιπτώσεις και στην επάρκεια της σύνταξης. Είχαμε πει ότι θέλαμε οι πτωχότεροι που ζουν κάτω από το όριο της ανέχειας να μπορέσουν να έχουν και αυτοί κάποια δικαιώματα. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Τι εξοικονομήσεις πρέπει να γίνουν. Και δεύτερον, για την ηλικία της συνταξιοδότησης. Συμφωνώ με όλους όσους λένε ότι δεν μπορούμε να καθορίσουμε μία πανενωσιακή ενιαία ηλικία συνταξιοδότηση. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει κάτι να κάνουν, κάτι να αποφασίσουν, να έχουν κάποια σύσταση. Ερωτώ λοιπόν τους πάντες το εξής. πώς θα, με τι τύπο θα τα εκφράσουμε όλα αυτά. Ξέρω ότι οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν τις απόψεις τους, αλλά πρέπει να το συνδυάσουμε. Και τρίτον, όλοι συζητήσαμε την οδηγία για τις συντάξεις και είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη έρευνα. Ερωτώ λοιπόν την Κομισιόν, τι σχέδια έχετε. Θα ήθελα να ξέρω τι αντιπροτάσεις έχετε. Γιατί νομίζω ότι η Κομισιόν θα δεχόταν κάποια αντιπρόταση. Μόνο τρία λεπτά μπορώ να σας δώσω. Όπως και τους υπόλοιπους. Η Business Europe. Ευχαριστώ. Καταρχήν υπάρχει το θέμα της ηλικίας συνταξιοδότησης και το ερώτημα του γιατί πάντοτε λέμε να αυξηθεί αντί να θέσουμε και το θέμα των χρόνων εργασίας. Από, για την Business Europe πρώτο βήμα μπορεί να είναι η αύξηση της ηλικία συνταξιοδότησης αλλά μετά από αυτό υπάρχουν και άλλα βήματα που μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό βέβαια εξαρτάται από, το, από την εθνική πραγματικότητα αλλά μπορεί να υπάρξουν και άλλοι μηχανισμοί προσαρμογής και θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα μπορούσε να καθοριστεί ένα περιθώριο όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν ορισμένες μειώσεις αν φύγουν νωρίτερα ή πριν αν φύγουν αργότερα κτλ για την καταπολέμηση της άνηση μεταχείρισης με βάση την ηλικία, ναι φυσικά δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο, αλλά ως εργοδότες εμείς το δεχόμαστε αυτό και ξέρουμε ότι πολλές εταιρείες προσπαθούν να πάρουν μέτρα καταπολέμησης της άνησης μεταχείρισης με βάση την ηλικία, ε, βελτίωση της ευημερίας στον τόπο εργασίας, αλλά και καθορισμό προγραμμάτων για να διασφαλιστεί ότι οι διαφορετικές ηλικίε των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη όπως πρέπει. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικό για μας να υπάρξει μια εξισορρόπηση μεταξύ παραγωγικότητας των εργαζομένων και κόστους τους. Και αυτό αφορά όλες τις ηλικίε για να είναι μια εταιρεία ανταγωνιστική. Ως προς τις άλλες ερωτήσεις που έχουν τεθεί, το θέμα της αναθεώρησης της οδηγίας ΙΟΡΠ έχει τεθεί αλλά νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή αναθεώρηση. Πρώτον γιατί έχει ήδη φέρει αποτελέσματα, όχι πολύ σημαντικά αλλά κάποια, και γενικά όταν μιλάμε για πιθανή αναθεώρηση της πρόβλημα θεωρείται η διαφορετική εφαρμογή ανακράτος μέλος. Αλλά επειδή είναι προβληματικός και ο ορισμός του τι θα ήταν μια διαμεθοριακή ή διεθνής εφαρμογή, θα έπρεπε πρώτα να τα αποσαφηνίσουμε αυτά και μετά να δούμε αν χρειάζονται αναθεώρηση. Τώρα η διαφοροποίηση των πόρων για τις συντάξεις. Πράγματι θα μπορούσαν να συνδυαστούν και, τα, και οι τρεις πυλώνες, αλλά και αυτό είναι θέμα των χωρών μελών. Για μας η διαφοροποίηση μεταξύ των τριών πυλώνων είναι ακριβώς ο καλύτερος τρόπος. Τέλος, για το αν χρειαζόμαστε πιο συστηματική η διευθέτηση σε ενωσιακό επίπεδο. Είχαμε ήδη πει ότι οι κανόνες που αφορούν τις πιτοχεύσεις όχι μόνο είναι ανεπαρκείς, αλλά θα, έχουν, θα είχαν επιπτώσεις και σε όλα τα συντεξιδοτικά συστήματα όλων των χωρών μελών. Ευχαριστώ ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα, αλλά σε μερικά. Μα λένε, μα γιατί μιλάτε συνέχεια για την ηλικία της συνταξιοδότησης. Γιατί αυτό το θέμα θέτει πέντε φορές η πράσινη βίβλος. Πέρα από αυτό όμως. να μιλάμε για παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης αλλά να μην μιλάμε για την πραγματική ηλικία όπου βγαίνει κανείς από το χώρο της εργασίας ή δεν έχει νόημα. Πρέπει να συνδυαστεί η πραγματική ηλικία της συνταξιοδότης με την νόμιμη ηλικία. Άλλο θέμα. είπατε να μην υπερκτιμούμε το δημογραφικό πρόβλημα. Πράγματι, αυτά είναι κυκλικά φαινόμενα που επανέρχονται και θα ήθελα να σας τονίσω το εξή. Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης τα καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης μετά τον πόλεμο εγκαθιδρύθηκαν σε εποχή που ήταν χειρότερη η δημογραφική κατάσταση. Και γιατί δημιουργήθηκαν, γιατί τότε υπήρχε απασχόληση και η ανοικοδόμηση. Γι' αυτό και μη συνδέουμε την ποιότητα της εργασίας και άρα πόρους για τις συντάξεις και συντάξεις. Η σύνδεση αυτή μας φαίνεται προφανέστατη, γι' αυτό επιμένουμε. Επίσης, έγινε λόγος για την ισότητα των φύλων τη στιγμή ιδίως της μεταξιοδότησης. Δεν μου αρέσει πολύ η αριθμητική, αλλά διαπιστώνουμε στην επαγγελματική ζωή ότι σήμερα οι μισθοί των γυναικών είναι χαμηλότεροι κατά 20% από τους μισθούς των ανδρών. Επομένως, στη σύνταξη πώς μπορεί να υπάρξει ισότητα. Πρέπει εκεί να δράσουμε κατά τη διάρκεια της ενεργού ζωής. Έπειτα. Αν πρέπει να φέρουμε, να μεταφέρουμε το βάρος στις επόμενες γενιές. Εγώ δεν μιλάω για βάρος, εγώ λέω ότι τα συστήματά μας λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε τουλάχιστον για το δημόσιο τομέα που είναι ο πιο ασφαλής και ο πιο αλληλέγγυος δείχνει ότι οι ενεργοί χρηματοδοτούν τη σύνταξη των συνταξιοδοτούντων. Εντάξει, αυτό είναι μια λογική από την οποία δεν πρέπει να βγούμε γιατί αλλιώς θα οδηγηθούμε σε καθαρά χρηματοπιστωτικά συστήματα που είναι ακόμη πιο επικίνδυνα. Δεν υπάρχει βέβαια θαυματουργή λύση, τη δέχομαι κυρία εισηγήτρια, αλλά να μην ξεχνάμε τα βασικά. Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμη, αλλά έχουμε μόνο τρία λεπτά κυρία Πρόεδρε και γι' αυτό ως συνδικαλιστής όλος ιδιαιτέρως θα είμαι επιθύνιος. Λοιπόν, ΟΑΠΕΜ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μου τέθηκε το συγκεκριμένο ερώτημα των προήμων συνταξιοδοτήσεων και της κατάχρησής τους. Ήταν αυτή η εύκολη λύση που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και κατά την κρίση, αλλά δεν είναι λύση αυτό. Εμείς ως εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν τη δεχόμαστε διαπιστώσαμε ότι οι πρώιμες συνταξιοδοτήσεις δεν επιτρέπουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας μία προς μία για τους νέους. Δεν είναι σωστό αυτό. Διαπιστώνουμε ότι όταν φύγει κανείς σε πρώιμη συνταξιοδότηση πολλές θέσεις εξαφανίζονται, δεν αντικαθίστανται από νέους. Αντίθετα, όσο πιο πολύ διατηρούνται οι θέσεις εργασίας, τόσο πιο πολύ μπαίνουν νέοι στην αγορά. Επομένως πρέπει να διατηρηθούν οι ηλικιωμένοι όσο το δυνατόν περισσότερο στον τόπο εργασίας. Παράλληλα δηλαδή να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης αλλά ιδιαίτερα η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης όπως είπε και ο εκπρόσωπος των συνουδικάτων. Και πρέπει να δράσουμε και για την κατάρτιση και για την παραγωγικότητα των μισθών και για την αύξηση τους που συνδέεται με την παραγωγικότητα και το κόστος. Να δοθούν κίνητρα φορολογικά, να διατηρηθεί η ευελιξία ώστε να υπάρχει η επιλογή να παραμείνει κανείς έστω τμηματικά στην εργασία και τμηματικά στην μερικά στη σύνταξη. Εδώ χρειάζονται και ανοτομίες. Η αλληλεγγύη των γενεών είναι κάτι ιδιαίτερα απαραίτητο, έτσι δουλεύουν τα συστήματά μας αλλά πρέπει επίσης να υπάρξει διαφοροποίηση των πυλώνων. Γι' αυτό μίλησα για πολυπυλωνική προσέγγιση. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και την ατομική ευθύνη που φέρει. Δεν αρκεί να υπάρχει ευθύνη μεταξύ των γενεών, αλλά και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ευχαριστώ. Ο πρόσωπος του Ευρωκάδρου κύριος Παριέτη. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τελικά, επειδή άκουσα τις ερωτήσεις στα Ιταλικά. Μίλησα για πλαίσιο και για μέθοδο. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει ένα πλαίσιο στόχων, κριτηρίων και αρχών. Η μέθοδος βεβαίως συνίσταται στο τι θα κάνουμε μετά. Δεν γίνεται στην Ευρώπη να αποφασίζουμε εξ ολοκλήρου για το τι θα κάνουν τα εθνικά συστήματα. Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε και να θεσπίσουμε μεθόδους όπου με τον κοινωνικό διάλογο μέσω και της ηθικής της Λισαβόνας θα μπορούσαμε να καλέσουμε τους κοινωνικούς εταίρους και τα θεσμικά όργανα να καθορίσουν το πώς θα εφαρμόσουν τους στόχους αυτούς και τα κριτήρια και τις αρχές όσον αφορά τα διάφορα εθνικά συστήματα, δημιουργώντας δηλαδή ένα σύνδεσμο που σήμερα δεν υπάρχει και τόσο μεταξύ διαλόγου σε ευρωπαϊκό και διαλόγου σε εθνικό επίπεδο. Για θέματα τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να αυξηθεί η συνολική ανταγωνιστικότητα του συστήματος και για να μειωθεί το κόστος της μη ή της έλλειψης εργασίας που το ευρωπαϊκό σύστημα σχετικά υψηλό. Θα μπορούσαν λοιπόν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ταυτόχρονα ευρωπαϊκές και εθνικές όσον αφορά τη συνεχή κατάρτιση. Ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να ξεπηραστεί η έλλειψη απασχόλησης στην ηλικία που ανέφερα προηγουμένως μεταξύ των 55 και 65 ετών. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να εφαρμόσουμε στις διάφορες καταστάσεις μέτρα που θα ήταν υπέρ των ίσων ευκαιριών ώστε να ξεπεράσουμε τις αδικίες και τις διακρίσεις λόγω φύλου που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Εδώ βεβαίως κάνουμε μια παραπομπή στο πλαίσιο και στη μέθοδο, δηλαδή να καθορίσουμε στόχους και να καθορίσουμε επίσης και μια μέθοδο που θα επιτρέψει την μεταφορά αυτών των στόχων σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο τελευταίος προσκεκλημένος κύριος Ανδρέας Τσίμερμαν. Ευχαριστώ θα αρχίσω απαντώντας στο ερώτημα ποιος θα πληρώσει για τις συντάξει στο μέλλον. Για μας το κλειδί της χρηματοδότησης βρίσκεται στην αγορά εργασίας. Είναι απαραίτητο να έρθουν να μπουν περισσότεροι στην εργασία. Και επειδή εκπροσωπώ μια οργάνωση που τα μέλη της έχουν πετύχει στη δουλειά τους, θα έλεγα ότι οι δουλειές που χρειαζόμαστε είναι ποιοτικές, γιατί χωρίς περισσότερη ειδικευμένη και υψηλή ποιότητα εργασία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι συνεντάξεις. Πράγμα που με οδηγεί και στο ερώτημα του ελεύθερου χρόνου και της ηλικία. Αν υπάρχει δηλαδή διαμάχη εδώ μεταξύ πιο ηλικιωμένων και νεωτέρων. Εδώ συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Βολοζίνσκι. Κατ' εμάς η πρώιμη συνταξιοδότηση έχει δημιουργήσει τεράστιο βάρος σε όλους τους εργαζόμενους, σε ολόκληρη την κοινωνία και τους νέους και τους μεγαλύτερους, χωρίς να βελτιώσει τις ευκαιρίες τους να μπουν στην αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να τα δοκιμάσουμε όλα και την παράταση της ηλικίας συνταξιοδότης και τα υπόλοιπα. Όσο για τη διαφορετική μεταχείριση των ηλικιών, αναμένουμε από την Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τις δικαιοδοσίες που έχει για να καταπολεμήσει την άνηση μεταχείριση των ηλικιών. Αυτό δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τους πιο ηλικιωμένους, αλλά πολλές φορές και τους νεότερους. Ιδιαίτερα ως προς τα κατώτατα όρια που απαιτούνται για συνταξιοδότηση. Τέταρτον, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Μαν για τη διατήρηση των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας που βοηθάει τα πράγματα. Όντως αν υπάρχει σταθερή εργασιακή σχέση και συμφωνία ότι η σχέση αυτή πρέπει να είναι διαρκής και συμφωνούν οι δύο πλευρές για την σταθερότητα χωρίς να επιβάλλεται στο ένα από τα δύο μέρη η ευελιξία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστούμε. Η συζήτηση ήταν πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας για τα δημόσια οικονομικά και για τις συντάξεις. Στο μέλλον, στη συνέχεια, 22 Νοεμβρίου η συζήτηση για το πρώτο σχέδιο έκθεσης και συζήτηση με ορισμένους άλλους εμπειρογνώμονες Ευχαριστώ πολύ τους σημερινούς μας προσκεκλημένους και ερχόμαστε τώρα στο σημείο 18. Πριν όμως, πριν όμως λέγω, ξέρει κανείς αν έχει έρθει η κυρία Μωρέν του του του του. Όχι. Γιατί δεν θέλω να τελειώσουμε πριν μιλήσουμε για το θέμα που θίξαμε στην αρχή, δηλαδή τις τροπολογίες στην έκθεση της κυρίας Τσίμερ. Μερικοί συντονιστέ δεν είχαν έρθει τη τελευταία φορά, την Πέμπτη. Ιδίω η κυρία Αντιπρόεδρος που είχε την καλοσύνη να μου το γνωστοποιήσει τον προτέρων, αλλά εκτός αν έχω παρανοήσει νομίζω ότι οι συντονιστές έχουν πάθει αμνησία διότι στη συνεδρίαση των συντονιστών είχαμε ρητά πει ότι η συμφωνία μεταξύ Επιτροπής Γυναικών και Επιτροπής Απασχόλησης αφορούσε την κατανομή των δικαιοδοσιών και των καθηκόντων. Το είχαμε γράψει σε επιστολή σε όλους τους κοιόδης και τους συντονιστές και αυτό ακριβώς είχε συζητηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Αυτό ήταν το θέμα. Το θυμάμαι πολύ καλά. Εκτός αν ήταν απόντες όλοι οι σκιώδεις, αλλά αυτό τι να κάνω. Είχαμε λοιπόν αποφασίσει ρητά ότι εμείς θα μιλούσαμε για την ανέχεια και η Επιτροπή Γυναικών για τις γυναίκες. Γυναίκες ανέχεια, ανέχεια γυναίκες. Λοιπόν, αφού υπάρχει μια σαφή συμφωνία γιατί να επανέλθω. Δεν επανέρχομαι. Και άρα το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες τροπολογίες που δεν αφορούν αυτήν την κατανομή τι είναι σε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες οι σκιώδεις τις έκαναν αυτές τις αθέμητες τροπολογίες. Τους παρακαλώ λοιπόν είτε να τις επανυποβάλλουν αλλά στις γυναίκες, στην Επιτροπή Γυναικών, όπου υπάρχει διορία μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, είτε να υποβάλουν προφορικές τροπολογίες, αλλά γραπτός, για να δούμε αν μπορούμε να τις δεχτούμε. Αλλά χωρίς να τις ξαναγράψουμε από την αρχή, όχι. Γραπτός αλλά όχι ολόκληρες. Και αυτά αγγλικά ή γαλλικά. Ο κύριος Σέρκας αλλά μόνο για ένα λεπτό. Ναι, είναι σαφές ότι για τα θέματα φτώχειας είναι η Επιτροπή μας και για τα θέματα γυναικών είναι γυναικών. Έτσι είχαμε πει στους συντονιστές και αυτό είναι λογικό. Το πρόβλημα όταν είναι όταν μπερδεύονται αυτά τα δύο θέματα και πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη τροπολογία. Οι συντονιστές δεν τήρησαν μία προς μία την αρχή αυτής της τροπολογίας. Ναι, ναι, θα συναντήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδες για να δούμε θα κάνουμε τροπολογίες. Ωραία. Να μας μένει παρά να καθορίσουμε την επόμενη συνεδρίαση όχι, 18, διάφορα. Δύο-τρεις κανόνες όμως να έχουμε. Δηλαδή, προθεσμία συγγραφής και προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών στην Επιτροπή Γυναικών. Προτείνω λοιπόν μια συνάντηση για να ξεκαθαρίσουμε τις ε, τροπολογίες, όχι όμως για να ξαναγράψουμε μία προς μία τις τροπολογίες. Έτσι συμφωνούμε. Σημείο 18 διάφορα. Ζητώ συγγνώμη από τους προσκεκλημένους μας για αυτή την καθυστέρηση όσον αφορά την μελέτη της Νέας Ποσπονδίας για την αλλαγή του κλίματος, τις νέες βιομηχανικές πολιτικές και τους τρόπους εξόδου από την, από Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι είναι επίμαχο το θέμα των συντάξεων ως συνδικαλιστής και ότι μας οδηγεί στο να δαπανίσουμε περισσότερο χρόνο θεσμικό σε αυτά τα θέματα. Να σας παρουσιάσω αυτή τη μελέτη για την οποία έχουμε διανέμει μια... ένα φυλάδιο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω και να είμαι σύντομο και θα πω τα εξή. Αυτή η μελέτη ακολούθησε μια πρώτη μελέτη που έγινε από την, Ευρω... από τη Συνοσπονδία Συνδικάτων μία μελέτη του 2007 που είχε μεγάλη απήχηση ε, στον Παγκοσμίο Οργανισμό Εργασίας και αλλού και μας επέτρεψε να καθορίσουμε κάποιες έννοιες όπως ε, τις έννοιες της μετάβασης και της ε, πρόορης σύνταξης. Ε, συγγνώμη, της, της πρόληψης, συγγνώμη, συγγνώμη. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με τις κλιματικές αλλαγές και τις ανισότητες σε διάφορες περιφέρειες του κόσμου. Αυτό μας επέτρεψε να έχουμε επαφές με μη κυβερνικού οργανισμού στα πλαίσια ενός συντονισμού που ονομάζεται Spring Alliance το οποίο περιλαμβάνει κοινωνικούς εταίρους, συνδικάτα, μη κυβερνικού οργανισμούς και είπαμε ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα της κλιματικής αλλαγής αν δεν ασχοληθούμε με τα θέματα κοινωνικά, τα θέματα των διακρίσεων και των ισοτήτων σε πάντως σε συνδυασμό με το περιβάλλον. Στη συνέχεια κάναμε τη μελέτη αυτή τα προβλήματα της βιομηχανικής στρατηγικής. Η μελέτη αυτή είναι μεγάλη και έγινε εις βάθος, ανατομέα, σε συνεργασία με τις συνομοσπονδίες μας και θα ήθελα μόνο να τονίσω κάποιες πτυχές της. Καταρχήν, η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα αποτελεί μια πραγματική πρόκληση. Θα πρέπει να προσμετρήσουμε το τι αποτελεί σημερινή και ευρενή πρόκληση όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή το σύνολο των νέων τεχνολογιών και η επένδυση στην έρευνα στα επόμενα χρόνια, τομέα θα γίνει σύμφωνα με αυτή την πρόκληση για τη μείωση των εκπομπών διοξείου του άθρακα. Δηλαδή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα που αφορά όλες τις πολιτικές με την ιδιαιτερότητα της απαραίτητης ε, διασύνδεσης με την απασχόληση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό που ονομάζουμε δηλαδή προληπτική διαχείριση της απασχόλησης και το θέμα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης που σχετίζεται με αυτό το θέμα της ε, κοινοτομίας και της έρευνας. Υπογραμμίσαμε λοιπόν κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Μία από αυτές τις γραμμές, όπως μας έδειξε η μελέτη ανατομέα, η μελέτη βεβαίως θα δείτε στο φυλάδιο ε, αφορούσε το, σύλλογο, το σύνολο συγγνώμη, του τομέα της ηλεκτρικής ε, ενέργειας, τη σύνδρομη μηχανία, Να το αύριο τη σελίδα μου, που το γράφει, που το γράφει, καμιά βλακεία, αφορούσε, αφορούσε τη χημική μηχανία τσιμέντο, χάλιβα, Μηχανία γυαλιού, ε, δηληστήρια, μηχανία ε, μονοτικά υλικά κλπ. κλπ. Από αυτούς λοιπόν τους διάφορους τομείς προσπαθήσαμε να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε. Πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να σας αναφέρω για το σύνολο της μελέτης ανεξαρτήτως τομέα είναι ότι τα προβλήματα παγκοσμίω είναι σημαντικά. Το θέμα της αύξησης αυτών των δραστηριοτήτων τα προβλήματα που συνδέονται με αυτή την αύξηση των δραστηριοτήτων παραμένουν σημαντικά και είναι σημαντικά, οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποιο θα είναι το είδος της απάντησης και η εξέλιξή της. Γιατί το λέω αυτό, επειδή πράγματι σήμερα υπάρχει ένα διακυβευόμενο πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και το οποίο αφορά την αυριανή ανάπτυξη του κόσμου. Οι εκτιμήσεις του ΑΣΑ λένε ότι το 2050, το 30, η Ευρώπη θα πάει στο 9% συμβολή στην ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα πρέπει η τεχνολογία να μας βοηθήσει σε αυτούς τους τομείς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ε, κινδύνους της ταχείας από βιομηχανοποίησης λόγω ακριβώς της αύξησης των εκπομπών του άνθρακα. Έχουμε και το θέμα των αναπτυσσομένων χωρών το οποίο συνδέεται άμεσα με τις εκπομπές του άνθρακα και να σας δώσω ένα παράδειγμα αρκετά απλό. Το τσιμέντο σήμερα εδώ και τρία χρόνια εισάγεται στην Ευρώπη. Το τσιμέντο λοιπόν παράγεται εκτός Ευρώπης, είναι ένα εμπόρευμα με χαμηλή προστιθέμενη αξία και μεταφέρεται σε πλοία. Δηλαδή η Ευρώπη εισάγει το δικό της το τσιμέντο. Και αυτό επειδή ακριβώς είναι αποκεντρωμένες οι κύριες αγορές τσιμέντου, και η μεγαλύτερη βιομηχανία στην Κίνα είναι η Λαφάρς. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα αξιοποίησης της ε, αποκέντρωσης μηχανικής και της μείωσης των εκπομπών διοξίου του άνθρακα. Και να πω επ' αυτού ότι οι διεθνικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις λένε ότι υπάρχει κίνδυνος βεβαίως για τον άνθρακα στην Ευρώπη, ταυτόχρονα όμως ανοίγουν κέντρα ερευνητικά σε όλες τις χώρες, τις αναπτυσσόμενες ιδιαίτερα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξή. Είδαμε και την ε, οικονομική κρίση και το κατά πόσο αυτή κατέδειξε τον υψηλό βαθμό χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα ή χρηματοοικονομικού χαρακτήρα της ανάπτυξης που είχαν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα να δώσουμε απαντήσεις μέσω έρευνας και καινοτομία που θα μας επιτρέψουν να εφαρμόσουμε πολιτικές μέσω μακροπρόθεσμες γιατί είμαστε σε μια έτσι κάπως ιδιαίωσα εβδομάδα τώρα επειδή η Κομισιόν θα ανακοινώσει την πρότασή τη για τη νέα αγορά για την βιομηχανική πολιτική στο μέλλον και τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες, νομίζω το Δεκέμβρη, θα έχουμε και ένα συμβούλιο για την ενέργεια και θα έχουμε τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την ενέργεια και την ενεργειακή πολιτική της Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το σύνολο των χρηματοοικονομικών πτυχών και την ικανότητα κλίμακος της Ένωσης να αντιμετωπίσει ακριβώς τα δικαιωμένα στον τομέα της έρευνας. Τη στιγμή που αυτοί οι τομείς βεβαίω έχουν ε, έντονη ενεργειακή απέτηση και χρειάζονται σημαντικές έρευνες. Θα πρέπει λοιπόν στην Ευρώπη να πάρουμε το παράδειγμα της ανακοίνωσης και να δούμε κατά πόσο το small is beautiful. Σε αυτόν τον τομέα το ύψος των επενδύσεων είναι σημαντικό. Δηλαδή βασιζόμαστε σε ένα τεχνολογικό φαινόμενο, τα κύματα, τα οποία ε, είναι κάτι το νέο και ε, είναι και δωρεάν. Δεν είχαμε τη δυνατότητα εδώ εφαρμογή συγκεκριμένων προτάσεων και λύσεων. Οπότε η απάντηση που θα πρέπει να δώσουμε στα ερωτήματα αυτά είναι μια απάντηση η οποία θα πρέπει να είναι μεγάλη εμβέλεια. Αν θέλουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα ανάπτυξη και διατήρηση τη οικονομία τη Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ακριβώ θα θέλαμε γρήγορα να καθορίσουμε τα τις τεχνολογικές δέσμες σε σχέση με τον άνθρακα θα πρέπει να ξεκινήσουμε συζήτηση στην Ευρώπη όσον αφορά την ύπαρξη μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας τυποποίησης και για τον κανονισμό REACH να πω ότι θα πρέπει να βρούμε την ανιχνευσιμότητα όσον αφορά τον άνθρακο, να διατηρήσουμε την ε, διεθνή ανταγωνιστικότητα. και για τη θέση των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων να πω ότι εμείς λάβαμε μία θέση όσον αφορά το ρίτς ανεχρησιμότητα και διαφάνεια είπαμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το θέμα no market no data, θεωρήσαμε ότι είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να μεταφέρουμε από την Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το REACH από αυτή την άποψη απαντούσε σε δύο ε, πτυχές, σε δύο αιτήματα, άνθρακας και τεχνολογία. Η διαδικασία όμως είναι μια διαδικασία, η διαδικασία του REACH είναι μια διαδικασία εκκίνησης, δηλαδή όσο θα βρισκόμαστε σε μια προχωρημένη τεχνολογικά κοινωνία, τόσο οι απαιτήσει ανιχνευσιμότητα θα είναι μεγαλύτερε για την οικονομία. Δηλαδή, οι κοινωνικέ ανισορροπίε και οι ανισορροπίε, οι φορολογικέ, δικαίου κτλ. θα είναι πάρα πολύ σημαντικέ μελλοντικά και οι συνθήκε τη αγορά θα επηρεάζονται από αυτέ τι ε, καταστάσει. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που αναφέρουμε λοιπόν στην μελέτη μα. Χρειαζόμαστε λοιπόν να κάνουμε κάτι για την έρευνα και την τεχνολογία, να επιταχύνω την παρουσίασή μου. Έχουμε όλα τα προβλήματα που σχετίζονται ε, με την ε, σύνδρομη μηχανία. Χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ κάποιες τεχνολογικές πλατφόρμες και την εξέλιξή τους. Χρειαζόμαστε ε, μια διατομιακή συνεργασία, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο όσον αφορά μάλιστα και τον άνθρακα. Για τον άνθρακα συγκεκριμένα έχουμε άλλο ένα κεφάλαιο αποθήκευση και συλλογή άνθρακα. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με την αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία αφιερώνουν εκατομμύρια δολάρια στην ανέβρεση και αποθήκευση άνθρακα και να πούμε ότι οι ενεργειακές ανάγκες είναι τεράστιες παγκοσμίως για να, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του πληθυσμού οπότε δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν ένα απόθεμα σημαντικό στην Ευρώπη επειδή η ανθρωπότητα δεν μπορεί να προβλέψει την ύπαρξη αποθέματος όσον αφορά τα αγαθά, θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια σημαντική ανάπτυξη στο σημαντικό πρόβλημα της αποθήκευσης του άνθρακα και μάλιστα η Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει σημαντικές έρευνες και έχουμε και κάποιες εμπειρίες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γερμανία, όμως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, το πρόβλημα της αποθήκευσης και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τη στιγμή που η χρήση των ορυκτών καυσίμων είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν κάποιε πτυχές πολύ σημαντικές εδώ. Μετά έχουμε και το θέμα της απασχόλησης και της έλλειψης ε, ανισοτήτων, της κατάργησης των ανισοτήτων. Είμαστε λοιπόν υπέρ και μάλιστα είχαμε και ένα ψήφισμα από αυτού στα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου άνθρακα. Είχαμε το θέμα που υποστηρίξαμε της αύξησης των ΑΠΕ, της ε, ενεργειακής απόδοσης και το θέμα των ε, μετασχηματισμών. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μία μετάβαση σωστή προς, ε, προς την ενέργεια. Θα πρέπει να έχουμε ποιοτικές θέσει εργασίας και αύξηση απασχόληση στην Ευρώπη. Δεν είναι βέβαια σίγουρο ότι θα έχουμε αύξηση της απασχόληση στην Ευρώπη από αυτού και να αναφερθώ σε δύο-τρία παραδείγματα. Η, η το κύριο μέρος ελληνική ελληνικών μορφών ενέργειας, η παραγωγή τους γίνεται στην ε, Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα τα οποία συνδέονται με την ενολική ενέργεια γιατί η, παραγωγή αυτών των στοιχείων, αυτών των στοιχείων που συνδέονται με την ενολική ενέργεια είναι τόσο επικίνδυνη που οι εργαζόμενοι δουλεύουν πάνω από τρεις εβδομάδες. Βεβαίω εμεί δεν έχουμε εμεί αρμοδιότητα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Φωτοβολταϊκά το ίδιο. Οι μπαταρίε των φωτοβολταϊκών παράγονται κυρίω στην Κίνα. Δηλαδή το κυριότερο κομμάτι, το μεγαλύτερο μέρο Παραγωγή ΑΠΕ γίνεται στην Κίνα, οπότε δεν ξέρει κανείς ακριβώς και πώ παράγονται. Έχουμε επίση και το πρόβλημα της, ε, των ε, εξειδικευμένων θέσεων εργασία και να σα δώσω άλλο ένα παράδειγμα για την ενεργειακή απόδοση. Η δημιουργία θέσεων εργασία όσον αφορά τον τομέα των κτηρίων ε, είναι πολύ σημαντική και είπα εδώ σε μια συνάντηση με τους πράσινους ότι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τα κτίρια σημαίνει ότι διασφαλίζουμε την τήρηση της διαφάνειας και των κανόνων όσον αφορά τους κανόνες εργασίας. Δηλαδή να μην έχουμε μαύρη εργασία, να μην έχουμε υπαπασχόληση, να μην έχουμε ε, ξέπλυμα χρήματος, να μην έχουμε διαφθορά. Οπότε η απέτηση για ύπαρξη ποιοτική εργασία σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντική και βεβαίως συνοδεύεται με τη φύση της εργασίας και τις συνθήκες και τους όρους της. Έχουμε λοιπόν ένα κοινωνικό διάλογο εδώ σημαντικό που πρέπει να γίνει και βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή όπου η Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες ανάπτυξης με ισορροπία, με διαφάνεια, με ανιχνευσιμότητα. Αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο ζητάμε από την Κομισιόν και θα κάνουμε συζητήσεις για αυτό το θέμα στα πλαίσια ενός ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου Τώρα βεβαίω και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε. Έχουμε και μια κοινή μελέτη με τους άλλους ε, κοινωνικού εταίρους, συνδικάτα και εργοδότες για αυτό το θέμα για την κλιματική αλλαγή και θεωρούμε ότι και τα θέματα της χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικά στο να διασφαλιστεί αυτή η μετάβαση προς την με διαχείριση, προς την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Ένα θέμα το οποίο μας φαίνεται σήμερα σημαντικό είναι το θέμα που αφορά τις θέσεις εργασίας. Δηλαδή το θέμα της διαφάνειας και της ανιχνευσιμότητα, αυτό που έλεγε και το Ρίτς, επειδή χρειαζόμαστε ακριβώς καλύτερη γνώση και μια καλύτερη ανάλυση αυτών των στοιχείων. Και στα πλαίσια πάντοτε του Ρίτς, το επίπεδο έρευνας όσον αφορά το πολλαπλασιασμό πολύπλοκων προϊόντων είναι ένα στοιχείο ουσιώδες που μας επιτρέπει να δούμε καλύτερα τις συνθήκες της ίδιας της εργασίας. Επειδή νομίζω ότι οι κλιματικές αλλαγές και η χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν γίνει πια ένα στοιχείο απαραίτητο της υγείας στον χώρο της εργασίας. Οπότε θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι επιταγές έχουμε και σε αυτό το τομέα. Για τις ΑΠΕ, τη βιοενέργεια, βιομάζα, για όλα αυτά βεβαίως είμαστε υπέρ της ανάπτυξής τους και βλέπουμε ότι στον τομέα της αυτοκινητομηχανίας ότι θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις όσον αφορά την εξέλιξη του τομέα αυτού και θα πρέπει να προβληθούν και κάποιες περίπλοκες μεταβατικές φάσεις όσον αφορά τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να προβλέψουμε δηλαδή μια μεταβατική φάση προ τα ευρυδικά αυτοκίνητα ή τα ηλεκτρικά, με κάποιε φάσει μεταβατικέ, οι οποίε όμω θα μπορούσαν να διαρκήσουν κάποια χρόνια, ώστε να παρανεύουμε κι εμείς τον τομέα της αυτοκίνησης όπου θα έχουμε σημαντικές μεταβολές στο μέλλον. Αλλά με υπόψη μας τώρα τον τομέα του άνθρακα η Ευρώπη θα πρέπει να γνωρίζει καλά την κατάσταση που επικρατεί στις διάφορες χώρες μέλη. Οι κλιματικές αλλαγές και ενέργεια το 2008 είχαμε μια υποεκτίμηση της μαρικής κατάστασης της ε, ενεργειακής ανάγκης της Ευρώπης όπως ε, για την περίπτωση της Πολωνίας. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η μορφή συνοχής που δίνουμε, ποια είναι η μορφή της πολιτικής βούλησης που έχουμε. Έναντι αυτών δεν πρέπει να ζητήσουμε από χώρα να παράγει 90%, που παράγει 90% της ε, ενεργειάς του από το άνθρακα να αναλάβει μόνο του την ευθύνη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναφερθούμε στην πρώτη συνθήκη της Ευρώπης, δηλαδή τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, όπου θα πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά την συνοχή και τις ε, χρηματοπιστωτικέ ενισχύσει. Αυτά είχα να σα πω. Η... Το έγγραφο, η προσούρα που έχουμε είναι πολύ πιο πλήρης από αυτά που σα είπα. Προσπάθησα να μην με μακρηγορήσω όμως και σα τα είπα πολύ σύντομα. No, euh, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή που είναι πάρα πολύ ουσιαστική για την εργασία τη δική μα επιτροπή γιατί μας ε, εντάσσει πραγματικά συζήτηση. Εγώ λυπούμαι που δεν είναι παρόντα όλα τα μέλη τη Επιτροπής μα για να ακούσουμε αυτή τη στρατηγική προσανατολισμού, την μέθοδο δηλαδή της ε, χρήσης των στοιχείων αυτών με τον τρόπο που μας τα παρουσιάσατε. Θα ξεπεράσουμε λίγο το χρόνο μας, αν μας επιτρέψουν οι διερμηνείς. Όχι πολύ. Η κυρία Σχέντερ και η κυρία Στάιμπρεκ μετά. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συμβολή σας αυτή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, όπω συζητήθηκαν και σημαντικά θέματα που αναφέρθηκαν, ιδίως το θέμα να υπάρχει κοινωνικό πλαίσιο για ένα διάλογο. Αυτό σχετίζεται πολύ συγκεκριμένα με τη δική μας απόφαση. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει εδώ ένα πολύ καλό παράδειγμα Λιόγκρινες που είναι στη ΣΥΠΑ όπου οι περιβαλλοντικές ενώσεις και οι και τα συνδικάτα προσπαθούν να συνεργαστούν για να βρουν μια λύση. Και υπάρχουν εδώ διάφορα στοιχεία συγκεκριμένα. Αυτό που είναι σημαντικό στην έκθεση επίσης είναι ότι εξετάσαμε πώς μπορούμε να ρωτηθούμε όχι μόνο στους νέους τομείς, αλλά και πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε τους, ε, τις αλλαγές, ιδίως όσον αφορά το θέμα της ε, εκπαίδευσης και μεταεκπαίδευσης, πώς μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο για να μην παραβλέψουμε τους εργαζόμενους και να μην απλώς παραμεριστούν. Μιλήσατε ε, για τομείς όπου γίνεται εντατική χρήση ενεργείας, εκεί η δραστηριότητα είναι διαφορετική, είναι ιδιαίτερη παραδείγματος χάρη στην Χαλιβουργία Το θέμα είναι πώς θα παραγάγουμε χάλιβα με λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και άρα μπορούμε να πούμε θα παραγάγουμε χάλιβα από αιωλική ενέργεια και άρα θα μειωθεί η κατανάλωση της ενέργειας και αυτό θα μπορούσε να προχωρήσει κι άλλο ακόμη. Και επίσης στην Γερμανία Κάναμε συζητήσεις με τα συνδικάτα και τι μας είπανε, μας είπανε ότι θα συνεχίσουν την νομοθετική διαδικασία. Όσον αφορά τα μέτρα αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας και ε, αυτό οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση της παραγωγής, πράγμα που καταδείχνει από την μετατροπή σε μία βιομηχανική κοινωνία πτωχή σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, έχουμε μεγάλο κέρδος. Και θέλω να αναφέρω επίση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης ένα κεντρικό θέμα της δικής μας έκθεσης, δηλαδή το δικαίωμα για μετεκπαίδευση, ούτως όλοι να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και ε, ευθύνη των συνδικάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Η κυρία Στάινμπρουκ και ποιος άλλο θέλει το λόγο. Φαίνεται όχι. Παρακαλώ κύριε Στάινμπρουκ. Ναι, σας ευχαριστώ. Μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που είπε η κυρία Σόντερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τα συνδικάτα και την ΕΤΟΥΚ για την έκθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητηθεί το θέμα ευρέως με όλε τι επιπτώσει και με όλες τι πτυχέ κάθε συγκεκριμένου τομέα. Στη δική μου περιφέρεια ε, υπάρχουν σημαντικέ επιπτώσει από τι αλλαγέ στη χημική και στην αυτοβιομηχανία και στην αυτοκινητοβιομηχανία και συμφωνούμε πολύ συχνά την σύγκρουση στόχων που <clears throat> απορρέουν από την εξέλιξη της βιομηχανικής πολιτικής. Είναι σημαντικό τα συνδικάτα να υψώσουν τη φωνή τους και να υποβάλουν προτάσεις για το πώς θα μπορούμε να κινηθούμε στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτή η διαδικασία αναδιάρθρωσης να συνοδεύεται και από τους εργαζόμενους, δηλαδή τα θέματα της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, κατάρτισης, καινούργιες απαιτήσει, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η σοσιαλιστική ομάδα εργάζεται έντονα πάνω στο θέμα αυτό και συζητάμε και ένα έγγραφο για πράσινες θέσεις απασχόλησης. Θα το υποβάλουμε αυτό το έγγραφο για να προωθήσουμε τη συνεργασία μας. Χρειαζόμαστε πράσινες θέσεις απασχόλησης. Και κατά τη γνώμη μου, οι συγκρούσεις των στόχων μπορούν να επιληθούν άμα διευρύνουμε κάπως τον ορίζοντα και άμα εξετάσουμε τις λεπτομέρειες. Αυτά γενικά και σα ευχαριστώ πολύ. Και σα ευχαριστώ. Τέσσερις παρατήρησει: Πρώτον, για την εμπλοκή της Κίνας εκεί μέσα εδώ υπάρχει καμιά φορά η αυταπάτη ότι είναι πολύ εύκολο να λυθεί το πρόβλημα με τη δημιουργία των πρασίνων θέσεων εργασίας, αλλά μπορεί να μην είναι ποιοτικέ οι θέσεις αυτές. γιατί το θέμα είναι τι κάνουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι δεν συμφωνούν μα, τόσο με, με, με τη διεθνή κοινότητα απλώς προσπαθούν να κερδίσουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και μάλιστα με συνθήκες που από κοινωνική ή περιβαλλοντική απόψεως μπορεί να είναι προβληματικές. Δεύτερον, η περιβαλλοντικη αποψεως μπορει να ειναι προβληματικέ. δευτερον η καταρτιση στην πραγματικότητα όχι τα μεγάλα ενεργειακά σχέδια, αλλά αυτά που λέμε για τις μεταρρυθμίσεις στα σπίτια, στη στέγαση, στις οικοδομές μπορεί να αφορούν μικρές επιχειρήσεις και επ' αυτού δεν υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πράγμα που δεν επιτρέπει και αδιαφορετικές χρηματοδοτήσεις. Τρίτον, η φορολόγηση του άνθρακος ή οι τιμές, οι τιμές του άνθρακα, του διοξιδίου δηλαδή. Δεν μιλάτε για ενεργειακή ασπίδα και αυτό με ανησυχεί. διότι για να αλλάξει ο κόσμος συμπεριφορά, για να φτάσουμε στο μείον 20% κατανάλωσης ενέργειας. Πρέπει να ξέρουμε ότι αν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας, τότε, τότε θα μειωθούν τα εισοδήματα των νοικοκυριών και δεν θα συμφωνεί αυτό καθόλου με την αρχή της προοδευτικής φορολόγησης γιατί τα φτωχότερα νοικοκυριά θα αντιμετωπίζουν την, τους ακριβότερους ενεργειακούς λογαριασμούς. Πώς λοιπόν μπορεί να συνδυαστεί αυτό το κίνητρο μέσω των τιμών χωρίς να δημιουργηθεί παράλληλα μια κοινωνική ανισότητα πολύ σημαντική. Ίσως αυτή η ιδέα της ενεργειακής ασπίδας να ήταν χρήσιμη. Τέλος, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σας θυμίσω τι έγινε με τα ανθρακοριχεία που δεν είναι ήταν τα πιο ανταγωνιστικά. Όχι εκείνα που συμφωνούν με το πρόγραμμά μας, αλλά εκείνα που γνωρίζαμε στη Γερμανία και την Ισπανία. όπου συζητήσαμε αν έπρεπε να συνεχίζουν να χορηγούνται εκεί επιχορηγήσεις κρατικές. Και το 14 προβλέπεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο το θέμα. Άλλες λένε, άλλα χώρες λένε το 18 να καταργηθούν οι επιχορηγήσεις αυτές και το Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας θέλει να το συζητήσει και αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Απαντήστε. Μάλιστα. Εγώ ευχαριστώ για τις ερωτήσεις λοιπόν. για την επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση. Στην πρώτη μελέτη μας για τις κλιματικές αλλαγές είχαμε πει ότι πράγματι πρέπει να υπάρξει μια κατάρτιση, αλλά το πρόβλημα εδώ που τίθεται, γιατί μιλήσατε για πράσινες θέσεις, είναι ότι δεν μπορούμε μέσω των πρασίνων θέσεων να δημιουργήσουμε πιο ασταθείς ακόμη συνθήκες εργασίας, γιατί είναι μεγάλος ο πειρασμός, πολύ μεγάλος. Και δεν πρέπει να αντιθέτουμε τις πράσινες θέσεις στις κίτρινες. Νομίζω ότι που λόγος. Νομίζω ότι σήμερα οι άμεσες επενδύσεις από έξω λαμβάνουν υπόψη τους το πρασίνισμα της βιομηχανίας και την τεχνολογική δυνατότητα του πρασινίσματος βέβαια οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτή τη στιγμή δεν, δεν ελέγχονται ακόμα. Αν κάποτε γίνει αυτό τότε καλά. Και τότε αυτό θα αφορά όλες τις θέσεις. Όλες. Γιατί υπάρχει εδώ ο κίνδυνος, ο πειρασμός να θεωρηθούν απαρχαιωμένες οι κανονικές θέσεις εργασίας μοντέ. Λοιπόν, ξέρω ότι ζούμε σε κοινωνία του marketing, αλλά δεν πρέπει να έχουμε αποτελέσματα αντίθετα από τα προσδοκόμενα. Λοιπόν, και γιατί το λέω, διότι, διότι να, όλες οι αφορούν. αφορούν. Αν πρασινίσουν όλες, τότε καλά. Και τότε αυτά θα γίνουν όλα οι αλλαγέ στην αγορά εργασία, θα γίνουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αλλά, αλλά με τη Βελγική Προεδρία και την Κομισιόν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πρόβλεψη των μεταρρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων, να δούμε τι μπορεί και πώς θα γίνει. Και πρέπει βέβαια να έχουμε ένα όραμα και κοινωνικό και κοινωνιακό. Για τις τιμές τώρα ή το τίμημα, τις τιμές, τις τιμές. Εδώ υπάρχει χωριστό ψηφίσμα, χωριστό για την ενέργεια, για τις τιμές. Ε, πρόκειται να οργανωθεί ένα συμβούλιο το Δεκέμβριο και στις 24 Φεβρουαρίου διάσκεψη των αρχηγών κρατών αλλά και κυβερνήσεων και Στι 24 Νοεμβρίου επίση άλλη διάσκεψη θα οργανώσουν η Βελγική Προεδρία για το θέμα των ενεργειακών τιμών για να μην ενδυναμωθούν οι ανισότητε μέσα στι χώρε γιατί η αύξηση των τιμών τη ενέργεια για τους πτωχότερους θα αποτελέσει πραγματικό πρόβλημα και η αποτελεσματική και οικονομικότερη χρήση μπορεί να δημιουργεί προβλήματα και άρα υπάρχει εδώ ένα θέμα οργάνωσης που το λένε ορισμένη ενεργειακή ασπίδα. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για όλα αυτά. Ποια είναι η σωστότερη τιμή της ενέργειας. Λοιπόν, για το θέμα του άνθρακος τώρα. Λοιπόν, του άνθρακος για τα μεταβατικά μέτρα καταρχήν, ως συνδικαλιστής θα τα πω. Λοιπόν, ε, όπως έλεγε ένας διάσημος Γάλλος πολιτικός, ε, που του λέγανε δεν είναι καλή αυτή η απάντηση, έλεγε ναι αλλά αυτή την απάντηση έχω να σε λοιπόν αυτό θα πω και εγώ λοιπόν. Για την Ισπανία ιδιαίτερα, στην Ισπανία που είναι τεταμένα τα πράγματα, η αγορά εργασίας είναι εύθραυστη και εκεί είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς. Ε γιατί οι αλλαγέ στην Ισπανία είναι πολύπλοκες και δεν μπορεί κανεί να τα δει πρόθεσμα. άρα μόνο μεσοπρόθεσμα και άνω. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν του άνθρακος, τι να σας πω, υπήρχε μια αρχική μέθοδος από την ΕΚΑΧ, τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλη μέθοδο, πιο σφαιρική, πιο... την είχαμε προτείνει πριν από λίγο. Χρειάζεται μια προσέγγιση που να είναι σαν τη ΕΚΑΧ, αν θέλουμε να υπάρξει συνέπεια, συνοχή και αλληλεγγύη. Αν δεν θέλουμε πιο αλληλέγγυα προσέγγιση, τότε, ξέρετε, με την προηγούμενη επιτροπή είχα συνεννοηθεί για το θέμα της ενέργειας και είχαμε διαπιστώσει ότι η αγορά του φυσικού αερίου δεν είναι κανονική αγορά γιατί υπάρχει δεσπόζουσα θέση του Γκάσπρομ και αυτό δημιουργεί προβλήματα στη Λιθουανία, στην Ισθονία. Είναι τεράστια προβλήματα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν εδώ κάποια επένδυση, δεν είναι μόνο το θέμα των καταρτήσεων, αλλά η έρευνα, η επένδυση είναι θέμα που τίθεται στην Ευρώπη και εδώ πρέπει να γίνουν αλλαγές στον ενεργειακό τομέα. Είναι επενδύσεις μέσω και μακροπρόθεσμες που δεν ενδιαφέρουν τις, τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Δεν θα ενδιαφέρει. Χρειάζονται λοιπόν μακροπρόθεσμα, μακρόπνοα προγράμματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για την απάντησή σας που θα μας εμπνεύσει οπωσδήποτε για τις μελλοντικές μας εργασίες. Θα τις συζητήσουμε μεταξύ μας να μπορούσαμε να προετοιμάσουμε τη δική μα θέση και το κοινό βιβλίο σε αυτό. Ολοκληρώσαμε τι εργασίε μα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα του διερμηνεί που μα έδωσαν λίγο χρόνο παραπάνω και θα τα ξαναπούμε στην συνεδρίασή μα στι 8 και 9 Νοεμβρίου.